Συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, έχουμε αργήσει, αλλά κόλλησε στην κίνηση ο κ. Σταγιάννη. Καμιά φορά, ξέρετε, είναι πιο εύκολο να πάει κανείς στο Ασβούργο από να έρθει εδώ πέρα από την Κομισιόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Επίτροπο που ήρθε να μας μιλήσει σήμερα και με μεγάλη μας χαρά σας έχουμε κοντά μας. Είδαμε τον ε, Μισελ Μπαρνιέ για το ίδιο θέμα πριν από ε, λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες και πάντα για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Άμυνας. Και συγκροτήσατε με τον κύριο Μπαρνιέ μια task force, περιμένουμε πώς και πώς σχετικές ανακοινώσεις όσον αφορά την βιομηχανία άμυνας. Είπα ότι θέλουμε να δούμε πώς θα γίνει αναδιάρθρωση, πώς θα αποκτήσει ανταγωνιστικότητα, πώς θα κινηθεί εμπορικά η βιομηχανία αυτή. Γιατί επ' αυτού επιδέχεται πολύ βελτίωση η κατάσταση μας πείτε επομένω τις δικές σας θέσεις, να μας πείτε τι γίνεται πλευράς κομισιών, τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Χθες είχαμε ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, μιλήσατε εσείς για τις θέματα άμυνας και οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι η συζήτηση έχει λάβει πολύ σοβαρό χαρακτήρα όσον αφορά την ακολουθητέα στρατηγική, δηλαδή μια βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμυνας που και εσείς προωθείτε. Μια ευρωπαϊκή τέτοια βιομηχανία. Να μας πείτε επομένω τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε, τι παραμέτρους, γιατί πρόκειται για ένα κλάδο που δεν είναι σαν τους άλλους. Έχει πολλές ιδιομορφίες, λόγω οργάνωσης, λόγω σκοπού, λόγω δυνατοτήτων που δίνει στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να έχουν δυνατότητες στρατιωτικής επέμβασης. Άρα, πρόκειται για νέο θέμα. Όλοι ενδιαφερόμαστε. Και βεβαίω με μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Θα σας δώσω τη σκητάλη και κατόπιν θα ακούσουμε τους συναδέλφους της υποπίτροπης. Αλλά και τους συναδέλφους με την Επιτροπή Βιομηχανίας που έχουν προσκληθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφαλείας και Αμήνης ως Επίτροπος, αλλά ήμουν παλιό μέλος της Επιτροπής αυτής όταν ήμουν Ευρωβουλευτής, οπότε είναι πάντα για μένα χαρά να παρίσταμαι εδώ και να είμαι ανάμεσά σας. Όπως είπατε, χτες συμμετείχα στην ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμήνης, όπου παρουσίασα τη στατική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν παρουσιάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν σώμα το κείμενο για τη βιομηχανική πολιτική άμυνας. Δεν θέλω την είναι κάστρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ, όπου οι επίτροποι και οι υπηρεσίες ετοιμάζουν ένα κείμενο ε, που θέλουν να το επιβάλλουν στους άλλους, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη θέση της πριν ετοιμάσει ένα κείμενο, όμως και υποβάλει στο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα κείμενο, πρέπει να παρουσιάσει ιδέες, να ακούσει τις τοποθετήσεις των διαφόρων θεμάτων και μετά να υπάρξει δυνατότητα συζήτησης ε, των θεμάτων και κυρίως για ένα ειδικό θέμα, όπως αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική αμήνης ε, θα υπάρξει αυτό το Συμβούλιο στο τέλο του έτου, θα πρέπει να υπάρχει βιομηχανία αμυντική. Εξήγησα γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να έχουμε βιομηχανική πολιτική ευρωπαϊκή αμήνη. Αυτό δεν σημαίνει να αλλάξουν οι κανόνε. Ή ε, ε, να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κάτι στα διάφορα κράτη-μέλη, πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τα πράγματα χωρί να αλλάξουμε του κανόνε τη επικουρικότητα. Να μην επιβάλλουμε κάτι αλλά πρέπει να υπάρχουν πρότυπα, να υπάρχει συντονισμένη βιομηχανική πολιτική, διότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε έτσι πολλά χρήματα και αυτά σε μια τέτοια κατάσταση κρίσης πρέπει να γίνει, θα πρέπει να έχουμε πρότυπα για να είναι πιο αποτελεσματική η δράση των στατευμάτων μας και στις ειρηνευτικέ επιχειρήσει και επιβολή τη ειρήνης. Peace δεν πρέπει να συμβούν ξανά αυτά που συνέβησαν ε, που συνέβησαν στην πρώην Κυκοσταβία κατά το παρελθόν, που είχαμε τα άρματα μάχη στον άλλο και δεν υπήρχε συνεννόηση. Ε, είχα θετική απάντηση. Τα κράτη-μέλη πάντα ανησυχούν. Θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλλει κανόνε όσον αφορά και την εθνική ασφάλεια. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να συντονίσω να έχουμε πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και ο τομέα τη αμυντική βιομηχανία είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό τομέα σε μια στρατηγική υπέρ της επαναβιομηχανοποίησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεω Έχουμε ποιοτική βιομηχανία, μπορούμε να κερδίσουμε την πρόκληση σε παγκόσμιο προσκήνιο και να προωθήσουμε την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Στην αμυντική βιομηχανία έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Το Συμβούλιο άκουσε Ζήτησα από τα κράτη-μέλη να στείλουν προτάσεις, ιδέες ε, πριν εγκριθεί το τελικό κείμενο και το ίδιο ζητώ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν έχετε ιδέες, έχετε προτάσεις ε, ας ε, ακουστούν. Μην διστάζετε, όχι μόνο σήμερα στη συζήτηση να εκφράσετε απόψεις, αλλά και στο γραφείο μου, το γραφείο μου, η υπηρεσία μου, είναι έτοιμοι όλοι να λάβουν προτάσεις, συστάσεις κλπ. Αφού ακούσατε και αυτά που είχα να πω που θα παρουσιάσετε στι Ευρωπαϊκέ Εγώ όμω μπορώ να σας ακούσω και να λάβω πληροφορίε, ιδέε, κλπ. Ό,τι σας ενδιαφέρει. Επί του θέματος, πριν την έγκριση του κειμένου, που πιστεύει ότι ο Επίτροπος Μπανία και εγώ θα προτείνουμε στο σώμα πριν το καλοκαίρι. Πριν σας εξηγήσω τι κάνουμε, δεν είναι κάτι αποφασισμένο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, διότι είμαστε ανοιχτοί στα όσα έχετε να πείτε, σας ακούσουμε. Θα ήθελα να πω και μερικά λόγια σχετικά με τη διαστημική πολιτική και να παρουσιάσω συνοπτικά τις εργασίες της Νέας Υόρκης για την συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Θα γυρίσω στην γλώσσα μου τη μητρική στα Ιταλικά. Σας είπα λοιπόν ότι το 2013 είναι μια χρονιά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, όχι μόνο διότι υπάρχει το Συμβούλιο, αλλά θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε όσον αφορά τη δράση που θα υποβάλει προτάσει. Η παρούσα κατάσταση έχει απαιτήσει όσον αφορά την ασφάλεια και απαιτήσει γίνονται όλο και πιο ε, μεγάλες. Και όπως είπα όμως προηγουμένως μειώνονται και οι πόροι. Άρα χρειάζονται κατεπίγουσες και κοινέ δράσεις. Δεν μπορούμε να βάλουμε αποφάσει όσον αφορά τι ανάγκε για το στρατιωτικό δυναμικό, διότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία του τομέα θα υποφέρει και όλα όσα, όλοι όσοι εξαρτώνται από αυτό και το έσοδό του. Είναι μεγάλο ο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα τη αμήνα και αυτό που είπα δέχτηκε πάρα πολλά θετικά σχόλια πλευρά των Υπουργών των διαφορών κρατομελών. Θεωρώ λοιπόν απόλυτα θετική την επιλογή του Συμβουλίου να αφιερώσει μια συζήτηση στο θέμα αυτό. Προφανώς αυτό το τμήμα της μηχανίας που μόνο το 2010 είχε τζίρο 94 δις ε, προσελκύει την καινοτομία και πολύ ψηλή τεχνολογία. Οι δραστηριότητε έρευνα και της ανάπτυξη στον τομέα τη άμυνα ε, αυτά ε, έχουν και συνέπειες και για άλλους τομείς όπως ηλεκτρονικά, το διάστημα και η πολιτική αεροπορία και οι στην άμυνα εν γέννη οδηγούν και σε δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασία που απαιτούν πολύ ψηλά προσόντα. Αν θέλει η Ευρώπη όμω να είναι πραγματικά να ηγηθεί στην καινοτομία και την έρευνα θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα αυτού του τομέα που είναι στατική σημασία και αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο τη βιομηχανική μα πολιτική που έχει σαν στόχο να πετέχει το 20% του ΑΕΠ της Ευρώπης που θα προέρχεται από την ε, βιομηχανία πριν από το 2020. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ενετόπισε τρία σημεία κλειδιά, τα οποία θα συζητηθούν το Δεκέμβριο. Πρώτα απ' όλα η ενίσχυση του δυναμικού της πολιτικής ασφαλείας και της κοινή άμυνας, δεύτερον βελτίωση της διαθεσιμότητας των διαφόρων αμυντικών μέσων και εργαλείων και τρίτον αυτό που είναι αρμοδιότητά μου και αρμοδιότητα του συναδέλφου μου του κυρίου Μπαρνιέ είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας η πολιτική της ασφάλειας και άμυνας, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, θα γίνουν αυτές οι πολιτικές αξιόπιστες αν υποστηρίζονται από μια ισχυρή στέρη βιομηχανική βάση που θα είναι σε θέση να δίνει εργαλεία και λύσεις που θα είναι αποτελεσματικές ταυτόχρονα ανταποκρινόμενες στις μελλοντικέ προκλήσεις και τις σημερινές. Η ανακοίνωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας που θα υποβάλουμε μαζί με τον Επίτροπο Μπαρνιέ θα επικεντρωθεί επί κάποιων ε, γραμμών δράσεως. Ε, πρώτα απ' όλα, ε, εδώ θα μιλήσω για το πώς θα σωματωθούν οι δύο οδηγίες στην ένωμη τάξη των κρατών μελών όσον αφορά τις μεταφοράς των αμυντικών προϊόντων και των διαδικασιών διαγωνισμών για προμήθεια στον τομέα της ασφάλειας. Θέλουμε σε όλα τα κράτη-μέλη να γίνουν αποδεκτά αυτά τα μέτρα και θα επαγρυπνούμε ώστε, και να ζητώντα μάλιστα την υποστήριξη των κυβερνήσεων ούτως ώστε να συμβεί αυτό εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν οι Και βέβαια και υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου όσον αφορά τα δύο νομοθετήματα που θεωρούμε σημαντικά. Ε, δεύτερο σημείο, όπως προανέφερα, που ήδη υποστηρίχθηκε αρκετά στο Συμβούλιο, αφορά το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, που κινδυνεύουν πολύ συχνά να υποφέρουν λόγω περικοπών ε, στις δαπάνες. Είναι δύσκολο έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντισταθμίσουν τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης με μια αύξηση των εξαγωγών προς άλλες χώρες. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε μέσω των κλώστες των συστάδων, των ομάδων, των επιχειρήσεων να υπάρξει πρόοδο στον τομέα τη αμυντική ε, βιομηχανία. Είναι ένα από του σημαντικού άξονε τη ανακοίνωσή μα. Τρίτο σημείο το οποίο υποστηρίχθηκε ευρέως από τους αμυντικούς φορείς Ευρωπαϊκής και από πλευρά του Συμβουλίου είναι και το θέμα της πιστοποίησης των αμυντικών προϊόντων. Μία εναρμονισμένη προσέγγιση για την πιστοποίηση των προϊόντων της άμυνας θα συνεπιφέρει σημαντικές οικονομίες, εξοικονομήσεις χρημάτων ε, και οικονομίες χρονικές και από πλευράς οικονομική. Θέλουμε να αυξήσουμε και τη δέσμευση Ευρωπαϊκή Υπηρεσία τη Άμυνα να κινηθεί και σωστά σε αυτό το τομέα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι των πρώτων υλών. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα και ξεχωριστά την άμυνα, αλλά ενδιαφέρει όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά και για την αμυντική βιομηχανία ε, πρόκειται περί ζητήματος ε, μεγάλης σημασίας. Άλλο σημείο είναι η σύμπραξη και η συνεργασία μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα. Καμιά φορά υπάρχει ιδεολογικός διαχωρισμός που, ε, που οδηγεί σε συμφορήσεις, να μην λειτουργεί καλά το σύστημα. Χρειάζεται ρεαλιστική προσέγγιση. Πρέπει να κινηθούμε με κάποια ευφυΐα ε, για να έχουμε καλύτερες, ε, να είναι υποφελής η προσέγγιση ε, και για το στρατιωτικό και το πολιτικό τομέα θα πρέπει να εντοπίσουμε και εκμεταλλευτούμε τους ιδιαίτερους τομείς που θα, θα επιτρέψουν, ε, θα αποφύγουν επικαλύψεις και να υπάρξει δυνατότητα επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και ε, τεχνολογική καινοτομία σε έναν ιό πλαίσιο πολιτικό και να υπάρχουν ταυτόχρονα θετικές επιπτώσεις και για τον πολιτικό και για το στρατιωτικό τομέα. Λοιπόν, Χρειάζεται διπλή κάλυψη. Χρειάζεται εξορθολογισμό και μεγιστοποίηση των επενδύσεων, αντισταθμίζοντα εν μέρη την μείωση των πόρων αυτές σε αυτή την περίοδο περικοπών των δαπανών και τη λιτότητα. Πώ μπορούμε δηλαδή να βελτιώσουμε την ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, λαμβάνοντα υπόψη τι συζητήσει που λάβουν χώρε όσον αφορά τον ορίζοντα 2020. Θέλουμε να προωθήσουμε υβριδικέ προδιαγραφέ για προϊόντα που μπορούν να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν και στον πολιτικό και στο δυτικό τομέα και προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική. Ένα άλλο τομέα, στον οποίο θα πρέπει, μπορούν να είναι μεγάλε οι ωφέλειε αμοιβέ, είναι ο τομέα του διαστήματο και των διαστημικών υποδομών και θα αναφερθώ εκτενέστερα αργότερα σε αυτό. Και τέλο, θα πρέπει να εξετάσουμε δελεχώστερα του τομεί στου οποίου η άμυνα και οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω έχουν κοινά συμφέροντα. Παραδείγματο χάρη, ενέργεια. Άλλο θέμα, το οποίο επιμακρών ε, συζητήθηκε χθε. Οι ένοπλε δυνάμει ευρωπαϊκέ έχουν μεγάλο συμφέρον και θέλουν να αλλάξουν ε, τον τρόπο κατανάλωση και την ποσότητα κατανάλωσης ε, των ε, καυσίμων των ορυκτών. Και γι' αυτό έχουμε σαν στόχο μέχρι το 2020 το στόχο 20-20-20 ε, για να ενισχύσουμε τη χρήση ανανεωσίμων πηγών ενέργεια και να μέσω κομπέ διοξιδίου του άνθρακο. Εν αυτή τη ενία βλέπουμε θετικό μάτι την θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Άμυνα που ε, ξεκίνησε το πρόγραμμα Go Green. Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό του πώς αυτοί οι στόχοι μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Λοιπόν, όπω έλεγα, η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εθετηθεί πριν από το καλοκαίρι, εξασφαλίζοντα χρόνο και χώρο για διαβουλεύσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επί τη βάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, θα ετοιμάσουμε ένα σχέδιο δράση λεπτομερέ για να υλοποιήσουμε τι διάφορε προτάσει και τι αποφάσει. Το θέμα τη αμυντική βιομηχανία και τη αμυντική πολιτική συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια τη συναντήσεω τη προπαρασκευαστική τη Λιθουανική Προεδρία, συνάντηση που υπήρξε μεταξύ Λιθουανική Κυβερνήσεω και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω γνωρίζετε, ο ίδιο ο Πρόεδρο Μπαρόζο σε πολλέ ομιλίε του υπογράμμισε πόσο είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό που συζητούμε σήμερα το απόγευμα. Εγώ θα ήθελα τελευταίες εξελίξεις για τη διαστημική μας πολιτική και όπως ξέρετε έχει και συνέπειες και αντίκτυπο αυτή η πολιτική για όλους ε, τους τομείς της ε, ασφάλειας. Ξεκινώντα από το Γαλιλαίο, Είναι η μεγαλύτερη υποδομή που είναι απόλυτα ευρωπαϊκή, εξ ευρωπαϊκή, που με τη θέση ισχύ στη λειτουργική φάση αυτού του προγράμματο, στο τέλο 2014, αρχέ 2015, θα ανοίξει μια τεράστια αγορά, νέα αγορά για πολιτικέ εφαρμογέ. Θα ήθελα να δραχτώ τη ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που έδωσε επί τη ευκαιρία των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του GNSS υποστήριξη που οδήγησε σε αυτή την πρωτοβουλία, που είναι η πρώτη πρόταση από το πακέτο ε, το, το πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, όπου κατέληξαν οι δύο συνομοθέτε σε πολιτική συμφωνία. Σημαντικό βήμα, που θεωρώ ότι είναι μια χειρονομία εμπιστοσύνη έναντι του Γαλιλαίου και του γεωστατικού συστήματο πλοήγηση του Ευρωπαϊκού, του ΕΓΝΟΣ. Αυτή η Επιτροπή έδειξε ενδιαφέρον για το Γαλιλαίο στην έκθεση της ε, Κόπα Ήδη το 2011 παρουσιάστηκε η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής αυτής όσον αφορά ε, τον ένα ρυθμισμένο δημόσια υπηρεσία. Ο δημικός μου στόχος είναι να παράσχουμε τις πρώτες υπηρεσίες από το τέλος του 2014. Θέλουμε να έχουμε 18 δορυφόρους εν χρήση μέχρι το τέλος αυτού του έτους και όχι λιγότερους από 26 μέχρι το 2016. Χτες μάλιστα έγινε μια συνεδρίαση με όλη τη συμμετοχή εκπροσώπων της ε, διαστημικής βιομηχανίας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο χρονισμός και οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν ήταν σωστές από πλευράς δημοσιονομικής. Λοιπόν, θα έχουμε από το νέο πολιτισμό πλαίσιο πόρους και έτσι θα αγοράσουμε τους, ε, τελικά και τους τόλους που απαιτηθούν δορυφόρων και των διαφόρων ε, χερσαίων εγκαταστάσεων που χρειάζονται και έτσι θα έχουμε ε, μια συστοιχία 30 ε, δορυφόρων ε, εγκαίρως. Για το Κοπέρνικος αποφάσισε να επανεντα... το Συμβούλιο στο Πολιτεύτη Δημοσιονομικών Πλαίσιο να επανενταχθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος Κοπέρνικος και αφορά την επιτήρηση και παρατήρηση ε, της γης Είμαι ικανοποιημένο διότι το Κοπέρνικου είναι σημαντικό. Εξασφαλίζει στην Ένωση να μπορεί να παρακολουθεί το περιβάλλον, εξασφαλίζει την ασφάλεια παράγοντας ε, ταυτόχρονα και θέσει εργασίας και ανάπτυξη. Ε, ξέρω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει ακόμα να εγκρίνει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά έχω την πεποίθηση ότι θα εγκριθούν και από αυτό το θεσμικό όργανο οι ε, αναγκαίοι πόροι. Όπω σίγουρα οι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια πρόταση για νέο κανονισμό για το Κοπέρνικο που θα πρέπει κανονικά να ευθετηθεί τι επόμενε εβδομάδε. Ζητώ την υποστήριξή σα για να πετύχουμε μια έγκριση γρήγορα, ώστε να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω την εφαρμογή του προγράμματο Κοπέρνικο, το οποίο νομική βάση εκπνέει το τέλο του έτου. Άλλο σημείο, οι υπηρεσίε εποπτεία ελέγχου του διαστήματος και ε, υπηρεσίες εντοπισμού. Δραστηριότητε τη εποπτεία του διαστήματο και εντοπισμού είναι βασικό εργαλείο που επιτρέπει στου χρήστε των δορυφόρων να μειώσουν του κινδύνου με αποτελεσματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιώντα λοιπόν για πρώτη φορά την ενομική βάση που αφιερώνεται στο διάστημα, πρότεινε ένα πρόγραμμα που προωθεί ε, μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εποπτείας Ελέγχου και Εντοπισμού Αυτά εδράζονται στους ήδη φυστάμενους πόρους που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, εγγυούμεθα έτσι και την επάρκεια των οικονομικών πόρων. Μπορώ να σας πω εκ των προτέρων ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εποπτείας και Εντοπισμού στο διάστημα θα είναι βασικό σημείο για την ανακοίνωσή μας για την άμυνα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πρακτική απόδειξη της σύμπραξης μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα. Το Κοινοβούλιο ζήτησε συχνά να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας του διαστήματο και ελέγχου του διαστήματο. Ε, είναι επιτάπητο η πρόταση και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στη βοήθειά σα. Λοιπόν, ξέρω και το επαναλαμβάνω ότι αυτές οι δραστηριότητες άπτονται στενά των εθνικών αμυντικών συμφερόντων και γι' αυτό θα πρέπει ε, να θα πρέπει να ενταχθούν οι εθνικοί πόροι στην υπηρεσία εποπτείας του διαστήματος στην Ευρωπαϊκή που θα είναι υπό τον έλεγχό του των εθνικών αρχών. Λοιπόν, για το εμπόριο όπλων τώρα, για τη σχετική συνθήκη που έχει συναυθεί. Ε, το παράνομο εμπόρια των συμβατικών όπλων ε, κοστίζει πάρα πολλέ ανθρώπινε ζωέ. Πάνω από 740.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά και οι γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο ε, από αυτά τα πτυχή αυτών των όπλων. Η διάσκεψη για τη συνθήκη για το εμπόριο των όπλων που έλαβε χώρα εδώ και ένα μήνα στη Νέα Υόρκη ήταν μια στιγμή μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε με τη δική της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τις εντολές που έδωσε το Συμβούλιο. Με χαρά σας ανακοινώνω σε τρει εβδομάδες Στι 2 Απριλίου, μάλλον, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων τη συνθήκη και στις 3 Ιουνίου που έρχεται θα θεθούν υπογραφές σε μια ειδική ε, τελετή. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα σχέδιο απόφασης που θα δίνει την άδεια στα κράτη-μέλη να υπογράψουν τη συνθήκη επί τη ευκαιρία της εν λόγω τελετής. Θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδε βήμα αυτό, διότι η συνθήκη θα καθορίζει προδιαγραφέ κοινέ δεσμευτικέ για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη μεταφορά συμβατικών όπλων το, το κείμενο της συνθήκης εμπεριέχει σαφείς διατάξεις όσον αφορά τη διαφάνεια και υψηλού επίπεδου προδιαγραφέ, καθώ και θέματα προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξασφαλίζει πέραν αυτών η συνθήκη ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογή που καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα όπλων συμπεριλαμβάνων των πυρομαχικών και άλλων ε, ανταλλακτικών. Πιστεύω ότι αυτή η συνθήκη θα συμβάλλει να καταστήσει το εμπόριο των όπλων κάτι πιο ε, υπεύθυνο και διαφανέ και είναι κοινό στόχο του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, μακρηγόρησα κάπω, όμω υπήρξαν πολλά πράγματα που ήθελα να σα πω, ε, διότι θα ήθελα το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί δεόντω επί όλων των πρωτοβουλειών, όλων των δραστηριοτήτων που μπορεί να ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας και πιστεύω ότι είναι σημαντικό εδώ να συζητηθεί το μέλλον της αμυντικής πολιτικής, της πολιτικής ασφάλειας και των συνεπειών που έχουν αυτές οι πολιτικές για την ε, ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής μας Ενώσεως. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, αγαπητέ Πρόεδρε. Αν υπάρχουν και άλλα σημεία προς διευκρίνηση, να σας δώσω τις αναγκαίες ε, πληροφορίες. Merci, monsieur Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, Διάφορες συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Να μην επιτρέπετε τις λεπτομέρειε για να το ξανασυζητήσουμε, αλλά θα ήθελα εγώ να σα υποπαρώ τι εξή δύο ερωτήσει. Και η Επιτροπή και τα κρατημέλη, από ό,τι φαίνεται, συζητούν τον προστατευτισμό. Λέξη που πολλές φορές προκαλεί θυμό. Και πρόκειται για κάποια πάρα πολύ ευαίσθητη σημαντική βιομηχανία όπως ε, η βιομηχανία της άμυνας με τις ιδιορυθμίες της. Τώρα όσον αφορά λοιπόν το εμπορικό, την εμπορική πτυχή αυτή της ε, ανακοίνωσης, αναφέρεστε εσείς στον προστατευτισμό. Πολλές φορές μιλάμε για αναδιάρθρωση, για ανταγωνιστικότητα και λέμε ότι μόνο οι δυνάμει τη αγορά μπορούν, μπορεί η αγορά τη δυνάμει τέλο πάντων να προσδώσει την αγωνιστικότητα σχεδόν αυτόματα. Μιλούμε για ευαίσθητε ε, τεχνολογίες, θέματα εθνική κυριαρχία. οπότε θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, λένε, προστασίας της τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Και ίδιε η ε, ΗΠΑ δεν απόκεινται μόνο στις δυνάμεις αγοράς. Έχουν και άλλα μέσα για να προστατεύσουν την βιομηχανία αμυνάς τους. Μας είπε ο Μισελ Μπαρνιέ. Ως παράδειγμα κάτι που είπε κάποιος υφυπουργό εμπορίου από την ε, Αμερική στο Μόναχο, ο οποίος χρησιμοποίησε τη λέξη προστασία που θέλει να χρησιμοποιήσει η, Αμερική για την αμυντική της βιομηχανία. Ποια είναι επομένω η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι θεωρητικό το θέμα. Σε αμέσως επόμενες εβδομάδες θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ πολιτικό και εξηγόντως πρακτικό. Για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις τώρα. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και πάντοτε επικαλείστε το ειδικό τους βάρος, τη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και στον τομέα της άμυνας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές φορές στριμώχνονται. Έχετε εσείς κάποια συγκεκριμένα μέσα, σχέδια τέλος πάντων για την προστασία των ΜΜΕ στον τομέα της άμυνας. Οπότε τώρα μπορούμε να αρχίσουμε τον γύρο τραπέζης. Ο κ. Λίζεκ, πρώτα-πρώτα, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεργαζόμαστε από καιρό, ε, κύριε Επίτροπε, και έχουμε και παρόμοιο τρόπο σκέπτεστε. Πολλά από αυτά που είπατε με βρίσκουν σύμφωνο. Νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούμε με την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής υποδομής. Άλλωστε, χρειαζόμαστε σύγχρονο εξοπλισμό. Και βέβαια εδώ παίζει ένα ρόλο και η κοινωνική πτυχή, η διασφάλιση της απασχόλησης στις χώρες μέλη της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί ειδικοί λέγουν ότι είναι αναπόφευκτο, γιατί σε περιόδους κρίσεως και παγκοσμιοποίησεως είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν ομαδοποιήσεις επιχειρήσεων, δηλαδή να συμπήξουν ομίλους πολλές μεσαίες, μικρές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό όσο αφορά κατασκευαστές αεροσκαφών, ε, πλοίων, ε, θωρακισμένων κλπ. Σε συνεργασία και με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι μειώνεται μεν ο αριθμός των κατασκευαστών, μεγαλώνουν όμως και σε όγκο και σε αξία οι παραγγελίες. Γι' αυτό και ρωτώ τον Επίτροπο πώς το βλέπει, ποια βήματα μελετά να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υποστηρίξουμε μάλλον τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ή θα δώσουμε μια μεγαλύτερη όθηση στη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και μήπως αυτό αποτελεί αντίφαση μεταξύ των δύο όρων. Και σε αυτά που είπε ο κ. Ντανζάν, εγώ συμφωνώ και τα υποστηρίζω. Αρχίζουν τώρα, αρχίζει ο σχεδιασμός των ε, διαβουλεύσεων για την μεγάλη διατλαντική αγορά μεταξύ Ενωμένων Πολιτιών και Ενωμένης Ευρώπης. Αυτά βέβαια είναι μελλοντικά οράματα αν θέλετε, αλλά μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα υπάρξουν και ότι θα καταργηθούν οι εμπορικοί φραγμοί. Πάλι εκεί οι ειδικοί μας λένε ότι αυτό ανοίγει πολλές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Μπορεί να αναλάβει παραγγελίες και για τον Αμερικανικό στρατό. Από την άλλη μεριά λένε ορισμένοι ότι αυτό σημαίνει και απειλή διότι σε ορισμένους τομείς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί και θα χάσουμε. Εσείς πώς το βλέπετε κύριε Επίτροπε. Η κυρία Κόπα παρακαλώ. Thank you, Mr. Commissioner. Ευχαριστώ Επίτροπε. Μια ισχυρή βιομηχανική βάση άμυνα είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των κρατών μελών και για τη φιλοδοξία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέα τη κοινή ασφαλεία και άμυνα. Και να υπάρξουν βήματα για νέα αγορά αμυντική είναι μια αναγκαιότητα. Ε, διότι είμαστε στο σημείο που θα πρέπει να ασχοληθούμε με το, τη φύση τη αγορά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό σε καλέ τιμέ για όλα τα κράτη-μέλη έχω να θέσω δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, πώ αντιμετωπίζεται το φαινόμενο τη διαφθοράς όσον αφορά τι δικασίες ε, προμηθειών. Το είπα αυτό διότι χώρε όπω η δική μου, η Ελλάδα, αλλά και άλλε χώρε, όπω είναι η Πορτογαλία που υποφέρουν τώρα από την οικονομική κρίση, έχουν εμπειρία τέτοιων φαινομένων, φαινομένων διαφθοράς ε, όσον αφορά τι προμήθειε. Και το συμπληρωματικό κόστο επιβαρύνει ε, όπως πάντα τους πολίτες. Το πρώτο ερώτημα είναι λοιπόν, ε, τι δες έχετε, σε ποιο βαθμό αυτή η Task Force εξετάζει το θέμα και μέτρα για την αντιμετώπιση των, ε, της διαφθοράς στο εμπόριο όπλων. Δεύτερον, ήδη εκφράσατε μια ιδέα, την ιδέα της αναδιάθρωσης της βιομηχανικής. Αυτό συμβαίνει και λόγω της οικονομικής κρίσης και αποτελεί και αναγκαιότητα διότι όπως είπε και ο πρόεδρος Ντανζάν, να ανταγωνίσουμε μια πιο καλή και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία στην απασχόληση και αν υπάρχουν μέτρα ή κατευθυντήριε γραμμέ που θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τα κατευθύρια κατά ε, κάτι μέρη να αντιμετωπίσουν τι κοινωνικέ συνέπειε ε, συγχωνεύσεων ή κλεισίματο μη βιωσίμων επιχειρήσεων είναι πολύ βασικό θέμα, ξέρετε, για την πολιτική μου ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Βανόρντεν. Um, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντώνιο, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω εδώ στην Επιτροπή. Στο τελευταίο αυτό που είπες για την συνθήκη για το εμπόριο όπλων, οι περισσότεροι από εμά είμαι σίγουρος καλωσορίζουμε αυτά που συνέβησαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστηρίζουμε ε, μια διεθνώς συμπεφωνημένη ε, συνθήκη για το εμπόριο όπλων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ε, θα σας ενδιαφέρει να σας πω ότι κατεβλήθη μια προσπάθεια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να ετοιμαστεί μια έκθεση που θα επέβαλε περισσότερους ελέγχους ε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάτι που δεν θα ήταν επικοδομητικό. Και σε ένα ξέσπασμα κοινή λογική, θα έλεγα, αυτό απερίφθη με 48 ψήφου έναντι μια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι ήταν, ε, αυτό που συνέβη ήταν άνευ προηγουμένου. Τώρα, επί της ουσίας. Και πάνω σε αυτά που μας είπατε, πολλοί από εμά θα προτιμούσαν μια πραγματιστική προσέγγιση όσον αφορά σημαντικές βιομηχανίες όπως είναι η αμυντική. Και θέλουμε ευρωπαϊκή εμπλοκή εκεί που υπάρχει προστιθέμενη αξία τι με προβληματίζει. Με προβληματίζει αυτό που άκουσα. Η φιλοδοξία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ΚΕΠΑ και κάποιοι πολύ θεωρητικοί στόχοι που τίθενται, σχεδόν θεολογικής φύσεω. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αμυντική βιομηχανία στις χώρες μας. Να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν το δυναμικό τους. Οι περισσότερε αμυντικέ μας ε, βιομηχανίε, συγκεντρώνονται σε πολύ λίγες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Έξι θα έλεγα. Έξι από αυτές έχουν πάνω από το 80% της ε, αμυντικής βιομηχανική παραγωγής. Και η έρευνα και η ανάπτυξη, η αμυντική συγκεντρώνονται σε ακόμα λιγότερες ε, χώρες. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείε έχουν συμφέροντα παγκόσμια εμβελίας αφήνοντας την BAE, η οποία έχει πολύ σημαντική ε, ε, παρουσία στις ΗΠΑ, η EADS έχει πάνω από 1,5 δις δολάρια τζίρο στη ΣΥΠΑ, η Τάλης πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια τζίρο στη ΣΥΠΑ, απασχολούν και οι δύο αυτές εταιρείες χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, είναι σαφές ότι στρέφουμε το βλέμμα εκτός Ευρώπης όταν μιλάμε για αυτές τις εταιρείε που σωστά ψάχνουν για αγορές, διασυνδέσεις και έτσι βγαίνουν εκτός Ευρώπης. Ε, αναφερθήκατε και στη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού. Αφήσατε να εννοηθεί αυτό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι είτε μέλη του ΝΑΤΟ ή κατά κάποιο τρόπο έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ ηγείται επί τυποποίησεως και διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού. Θα έλεγα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό σε σχέση με, τη, με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι ρόλος αυτός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα. Αυτά τα πράγματα ήδη ρυθμίζονται, γίνονται και δεν πρέπει να τα γνωρούμε. Άρα, πιστεύω και θεωρώ ότι το ερώτημα και το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώ μπορούμε καλύτερα να δώσουμε δυνατότητα σε ευρωπαϊκέ αμυντικέ εταιρείε να αναπτυχθούν και να πλουτίσουν μακροπρόθεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που είπατε για κοινή τυποποίηση και ε, τον, ε, του εξοπλισμού θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Ε, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να αφαιρέσουμε το στοιχείο της φιλοδοξίας από την εξουσία που δυστυχώς καθοδηγεί τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν. Η κυρία Λούζινγκ. Πρώτα-πρώτα και για να μην υπάρξει καμία παρανόηση, θέλω να πω ότι η επιρροή της ε, αμυντικής βιομηχανίας στην απασχόληση είναι σαφώς υπερτιμημένη. Μία ερώτηση τώρα για τις Προτινόμενε αναδιαρθρώσεις στην βιομηχανία όπλων που τα είπε και ο κύριος Λίζεκ ότι θεωρεί αναγκαίο να στηριχθούν κάποιες διαδικασίες συγχωνεύσεων, συγκεντρώσεων, το ίδιο φαίνεται να βλέπει και η Κομισιόν. Εγώ θέλω εκεί να σας θέσω το ερώτημα. Στη βάση ποιων μελετών ή άλλων πορισμάτων καταλήγεται στο συμπέρασμα ότι και άλλες παραπέρα διαδικασίες συγκέντρωσης θα μειώσουν το κόστος των αμοιβών στην βιομηχανία όπλων. Υπάρχει από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο μία μελέτη στις Ενωμένε Πολιτείε όπου η συγκέντρωση των βιομηχανιών όπλων είναι πολύ εντονότερη, διόλου δεν έχει οδηγήσει σε μείωση του μέσου κόστους εργασίας. Δεν αποδείχνεται κάτι τέτοιο. Και έχω και μια ερώτηση από τη δική σας σκοπιά. Πώς θα διαμορφωθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Θα μπει στην διακυβερνητική συνεργασία. Πώς θα ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου εφόσον η Κομισιόν στο μέλλον θέλει να παίξει ίδια μεγαλύτερο ρόλο. Και για την παρατήρησή σας για τον έλεγχο των εξαγωγών εξοπλισμών. Εγώ την παρακολούθησα με προσοχή και απαντώ σε αυτό που είπε ο κύριος Βανόρντεν, διότι εγώ το θεωρώ τουλάχιστον αξιοπερίεργο και διδάσκομαι, διότι συμβιβασμοί στους οποίους είχαν καταλήξει όλες οι πολιτικές ομάδες, όταν έρχονται να ψηφιστούν στην ε, Επιτροπή, φαίνεται ξαφνικά να αντιβαίνουν στην common sense. Εγώ νομίζω ότι μάλλον χρειάζεται, μάλλον γίνεται μια προσπάθεια να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε συζήτηση στην Ολομέλεια για τα θέματα αυτά. Πρώτη από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Ταϊάννη για την παρουσία σας που πάντα εκτιμάτε πολύ. Ξεκινώ από μια σκέψη. Η αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι πολύ κατακαιρματισμένη και θα έλεγα πολύ λίγο ανταγωνιστική. Η ίδια η άμυνα εξάλλου. Μιλάμε τα στοιχεία τα ίδια. Δύο εκατομμύρια άτομα είναι σε ένοπλε δυνάμεις συνολικά στην Ευρώπη. Στη ΣΥΠΑ 1,2 εκατομμύρια είναι στο στρατό, είναι στατευμένοι. Βλέπετε πόσο κατακαιρματισμένη είναι η κατάσταση και πόσο χαμηλή είναι η αποδοτικότητα όσον αφορά τον τομέα αυτό και τη βιομηχανία. Έχουμε ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αναφερθεί, της ε, πολιτικής αεροπορίας. Εκεί εφαρμόζεται σημαντική προσπάθεια σύγκλησης. Έχουμε την Airbus που είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε, πιστεύω, να πούμε το ίδιο για την αμυντική βιομηχανία μας. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με ένα συντονισμό. Με συντονισμό των δημοσίων αγορών, των, δημοσίων προμηθειών. Θα μπορούσε εντός του ΝΑΤΟ να υπάρχει δυνατότητα θεμητού ανταγωνισμού μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε τη βιομηχανία μας προς διαστάσεις μεγαλύτερες και μεγαλύτερο δυναμικό και αποτελεσματικότητα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όλη την αλυσίδα ε, προμήθειας, supply chain. Εκεί εμπλέκονται περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα μπορούσε να γίνει και σωστός εξορθολογισμός. Και αυτό θα ήταν αποφασιστική σημασία. Πιστεύω λοιπόν ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της άμυνας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι η διτή χρήση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια πραγματικότητα. Υποδομές, εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την στρατιωτική επιμελητεία αλλά και για την και για φυσικές καταστροφές. για την επιμελητία, για ε, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και για δημόσια χρήση. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό μάλιστα. Και λέω ότι αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη. Και για κοινές, σε πλαίσια κοινών ασκήσεων, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών να είμαστε πιο έτοιμοι, αν υπάρχει συνεργασία πολιτικού και εξωτικού τομέα. Πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα θέματα λεπτομερέστερα. Να καταφέρουμε να συγκλίνουμε την ευρωπαϊκή μας άμυνα, η βιομηχανία μας να γίνει πραγματικά ευρωπαϊκή, η αμυντική, και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους άλλους ε, κατασκευαστές με τους οποίους βεβαίως μπορούμε να μοιραστούμε ε, υποδομές και ίσως και σε κάποιες φάσεις και κάποια βέστητα μυστικά. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Τρεις ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων από πλευρά πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται εδώ και από του τρει βουλευτέ που ήθελαν να μιλήσουν, ο κ. Αγκουράκη, η κ. Ανιέ και ο κ. Τάνοκ. Μετά θα σα δώσω το λόγο για ένα τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Κύριε Επίτροπε. Πρώτα πρώτα θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη θέση μας. Εγώ υποστηρίζω 100% την επικουρικότητα. Α, δεν είναι εδώ να τα ακούσει ο κ. Φανόρνταν. Α, είναι ο κ. Στάνοκ, το ίδιο είναι. Οπότε, δεν θέλουμε ως Επιτροπή να αντικαταστήσουμε, να υποκαταστήσουμε τέλος πάντων τα κράτη-μέλη στον ρόλο το οποίο ε, παίζουν ε, για αυτές τις υποθέσεις. Αλλά όπως είπαμε και χθε στο Συμβούλιο, θα πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη μια προσθεμένη αξία. Δηλαδή, να κάτι το οποίο βοηθά τις οικονομίες, ε, την, ε, την άμυνα, σε όλα αυτά να κάνουμε περισσότερο. Κάτι παραπάνω, δηλαδή ποτέ δεν κάνουμε κάτι για να υποκαταστήσουμε τα κράτη-μέλη. Επίσης όσον αφορά την τυποποίηση, πρώτη υποποίηση, είπαμε στο κείμενο, αυτό το κάνουμε όταν ζητούν τα κράτη-μέλη από την Επιτροπή να οργανώσει, να προβλέψει, να καθιερώσει νέα στάνταρ νέα πρότυπα και, και σε νέους τομείς. Δεν το επιβάλλουμε. Εάν μόνο το ζητούν τα κράτη-μέλη. Το κάνουμε ούτω ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και όπως είπε ο κ. Βανόρδεν, όντως στο επίπεδο του ΝΑΤΟ ήδη υπάρχουν κάποια πρότυπα, αλλά εκεί δεν λειτουργεί δυστυχώς το σύστημα. Και οι πρωτοβουλίε δεν είναι πρωτοβουλίε του ΝΑΤΟ, είναι πρωτοβουλίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι δράσει ε, τη ε, ε, συμβολή τη ειρήνη, ε, οι ενευτικέ αποστολέ, οι δράσει κατά τη πειρατεία. Αυτά. Με την Ατλάντα έχουν σχέση περισσότερο. Άρα, θα πρέπει να γίνονται βήματα προ τα εμπρό. Δεν ξέρω, ίσως δεν, δεν το εξήγησα καλά ή δεν μεταφράστηκε καλά. Δεν μίλησα για συγκέντρωση, μίλησα για συνεργασία έτερων εκάτερων όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται να επιβάλλουμε συγκέντρωση. Μιλώ για συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Για να σου πω για τις ΜΜΕ για να απαντήσω και στη δεύτερη ερώτηση του Πρόεδρου. Θέλουμε να τις βοηθήσουμε. Το είπε και ο κύριος Λίζικ. Μία λύση είναι να μεγαλώσουν αυτές οι ΜΜΕ. Αλλά, όπως έχουμε κάνει και σε άλλους τομείς, μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα κλάστερ, τις συστάδες, του κόμβους. Να, και για τα πανεπιστήμια, όσον αφορά την έρευνα. Να, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό το έργο αυτό, το οποίο αφορά τις ΜΜΕ. Υπάρχουν λύσεις. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ είμαι υπέρ του να υπάρξει εμπορική συμφωνία, όπως είπαμε. Κατόπιν διαπραγματεύσεων θα πρέπει πάντοτε να είμαστε ε, έτοιμοι να σεβαστούμε τον θεμητό ανταγωνισμό. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για τους ευρωπαϊκούς Ευρωπαίους προμηθευτές προς τη ΣΥΠΑ. Το 12% ε, πιο πολλά ε, δίνουμε παρά παίρνουμε από τη ΣΥΠΑ. Είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα η αγορά αυτή. Γι' αυτό και στις ομιλίες με τη ΣΥΠΑ πρέπει να προσπαθήσουμε να μην υπάρχει προστατευτισμός, αλλά να γίνεται με όρους ισότητος η συνεννόηση. Μην είμαστε αφελείς. Κάποιοι όταν το λέω αυτό, θυμώνουν. Ε, καλά, λέω τότε δεν λέω αφελείς, λέω απλοϊκή. Αλλά οι μισέ από τι αμερικανικέ αγωγέ έρχονται από την Ευρώπη, λένε. Εντάξει, Α είμαστε προσεκτικοί, αλλά μην είμαστε αφελείς. Πάλι για τις ΜΜΕ. Καταβάλλεται προσπάθεια, να υπάρξει εναρμόνιση, να βοηθηθούν οι ΜΜΕ, να είναι πιο ανταγωνιστικές. Αυτά δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Μπορούμε να τις βοηθήσουμε, μπορούμε να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν και ταυτόχρονα μπορούμε να τις υπερασπιστούμε προσπαθώντας να τις εντάξουμε στο πλαίσιο, στη διάσταση των κόμμων των, των δεσμών, των κλάστερς. Δεν υπάρχει αντίθεση, αντίφαση. Τώρα όσον αφορά τη διαφθορά, όσον αφορά τις δισεκρατικές προμήθειες, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά πρέπει να γίνεται ορθή εφαρμογή των οδηγιών των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου που βοηθούν για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με όλα αυτά συμφωνώ. Να προσθέσω και κάτι άλλο για τον φίλο Βανόρντεν για την προτυποποίηση. Ναι, η Ευρώπη να αποτελεί προσθεμένη αξία και εγώ πιστεύω το ίδιο με εκείνον. Χθε, επίση, στο Συμβούλιο τη Άμυνα το είπαμε. Αλλά και η διαλειτουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είπαμε στο κείμενο τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προτυποποίηση. Λέμε για προτυποποίηση μόνο εάν το ζητούν τα κράτη-μέλη. προβαίνουμε σε προτυποποίηση μόνο αν μας ζητηθεί. Δεν θέλω τίποτε να επιβάλλω. Δεν ε, είμαι γραφειοκράτης. Δεν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια γραφειοκρατία. Την προτυποποίηση σας επαναλαμβάνω. Ενεργούμε μόνο όταν το ζητούν τα κρατημέλη. Λένε, μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε στους νέους τομείς νέα πρότυπα. Μόνο τότε ενεργούμε. Και συμφωνούμε τα όσα είπε ο κύριο Πρόντι για το κόστος της άμυνας. Δυστυχώ στην Ευρώπη το 51% του προπολογισμού καλύπτει το προσωπικό, ενώ είναι το αντίθετο στη ΣΥΠΑ. Πάνω από 20% πολύ λιγότερο από ό,τι δίνουμε εμεί. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε Πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα που διατίθενται για την άμυνα, μια που είναι τόσο σημαντικό τομέα. Και μπορεί να δημιουργηθούν νέες θέσει εργασία. Τώρα, όσον αφορά την αναδιάρθρωση, και την αναδιάρθρωση στους ευημέρους τομείς της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Έχουμε διάφορες ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, τα Διευθυντικά ταμεία, έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε την εργασία, τις τέσσερις εργασίας. Να προσπαθήσουμε να έχουμε στρατηγική για την προστασία της εργασίας και αυτό και κάνουμε με τον ε, Επίτροπο Αντόρ. να χαράσουμε μια στρατηγική. Τώρα, όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο, επίση και με το ταμείο αυτό υπάρχει συνεργασία. Je pense d'avoir répondu à presque toutes les questions. Νομίζω ότι κάλυψα όλε τι ερωτήσει. Α, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κάτι που το οποίο ανέφερε ο κύριο Πρόντι. Pourquoi la, la, la communication de la Commission Si nous voulons plus de compétitivité. Εάν θέλουμε περισσότερο ανταγωνιστική την βιομηχανία της άμυνας, θα πρέπει να αυξήσουμε τον συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαίων. Το, είπε ο κύριος Λίζεκ. Ε, ένα, κατάλογο με τις επιχειρήσεις. Αυτά ήδη τα έχουν κάνει και με το παραπάνω Αμερικανοί. Συντονισμός επομένως και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε οικονόμηση δαπανών, αλλά και η υπόθεση των προτύπων είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία. Δεν θέλουμε να γίνει κεντροκατευθυνόμενη. Να συγκρατηθεί το κόστος. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επίσης ε, Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Πρόεδρος. Καθυστερήσαμε για τον επόμενο κύριο ερωτήσεων. Κύριε Γιάννης, πρώτος εσείς, παρακαλώ όλοι να είστε σύντομοι. Γιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε κύριε Ταγιάννη για όσα είπατε που ήρθατε να μας δείτε και όπως είπαμε και στον κύριο Μπαρνιέ τα συγχαρητήρια έχουν να κάνουν με αυτή την θετική κατεξοχήν ευρωπαϊκή ιδέα της πρωτοβουλία που αναλάβατε να συγκροτήσετε αυτή την task force για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση στην βιομηχανία της άμυνας. Για να δούμε πώ θα έχουμε μια ευρωπαϊκή τέτοια βιομηχανία που να αντικατοπτρίζει την ουσία την ονομασία τη. Πολλέ φορές έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα για τις εθνικές ομοδιότητες και την υπηκορικότητα. Όχι, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο κόμπλεξ. Πρέπει να γίνονται βήματα προ τα εμπρό. Κάποια πράγματα με το περνάει χρόνος γίνονται απαρχαιωμένα, περιπίπτουν σε αχρησία. Μερικά πράγματα είναι αυτονόητο, δεν χρειάζονται εξηγήσει και επεξηγήσει. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι τι αποτελεί φραγμό, τι αποτελεί τροχοπέδι στην πορεία της Ευρώπης. Σας λέω πολλές φορές αυτό προκαλεί μελαγχολία να το σκέφτομαι. να λέμε για τεχνολογία χωρίς στοιχεία, για, για εξοικονόμηση δαπανών, για, για, διατήρηση της ειρήνης. Ναι, όλα αυτά μπορούν να αποκτήσουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα και να ξεκινήσουμε από την ε, βιομηχανία της άμυνας. Τότε σίγουρα τα πράγματα θα βελτιωθούν. Φυσικά και το τέλειο είναι να είμαστε μέσω αποτελεσματικοί σε όλους τους τομείς. Καλά, ε, ε, έχουμε και το φαινόμενο του προστατευτισμού, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί όπως οι άλλη κλάδοι της βιομηχανίας μας, και αυτός ο κλάδος της βιομηχανίας μπορεί να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους. Τους ανταγωνιστές της δηλαδή. Λέμε ξανά και ξανά για τον ΝΑΤΟ αυτά επιδέχονται συνεργασία και συμπληρωματικότητα. Και επίσης είπα είναι εταίρος, είναι φίλη χώρα, αλλά φυσικά και εκείνοι όπως και εμείς προσπαθούμε να πουλήσουμε περισσότερο και φυσικά είμαστε σε ανταγωνισμό. Όμως να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες του παιχνιδιού που να μην είναι υπέρ του ενός αλλά ούτε και υπέρ του άλλου. Δεν, είναι εδώ το θέμα είναι πώς θα βοηθήσουμε την βιομηχανία την ευρωπαϊκή. Είναι θέμα φιλοαμερικανισμού ή το αντίθετο. Αυτά πρόεδρε και ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Τσάλ Τάνοκ. Ευχαριστώ το ΝΑΤΟ. Δεν είναι απλώς ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι και πολλά κράτη μέσα Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Πολύ ευαίσθητο τομέα και επίτροπε εν μέρη απαντήσατε στο ερώτημά μου. Δηλαδή, το σώμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι άποψη έχει όσον αφορά τον πολύ ευαίσθητο τομέα τη εθνική κυριαρχία, δηλαδή τι ε, αμυντικέ προμήθειε. Όσον αφορά τι επικείμενε διαπραγματεύσει για το ΤΑΦΤΑ, δηλαδή χώρο ελευθέρου εμπορίου με τη ΣΥΠΑ, που ελπίζουμε να λάβει χώρα. Το όλο θέμα ε, ε, πολύ από τον Βρετανικό τύπο όταν η ADS πήγε να συγχωνευτεί με την BAE έπρεπε να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία του στατιωτικού βιομηχανικού τομέα και με το Υπουργείο Αμήνης των ΗΠΑ με την BAE και κυρίως στον τομέα των πυράβλων, πυραυλική συνεργασία στον τομέα των πυράβλων. Και δεν είπαν σχέσεις ε, ίδιες ε, μεταξύ Βρετανίας, είπα, όπως μεταξύ Γαλλίας, είπα, Γερμανίας, είπα και ούτω καθεξής πρέπει να ακολουθήσουμε συνεχτική προσέγγιση. Υπάρχουν δυνάμεις αγοράς. Λιτότητα στα εθνικά κονδύλια, τα αμυντικά κονδύλια. Και το ΙΠΑ μιλάει για αμαδοποίηση και μοίρασμα και ευφυή άμυνα. Και η ΚΕΠΑ μιλά για μοίρασμα της προσπαθίας. Και σιγά σιγά απομακρύνονται είπα, από την Ευρώπη, κινούνται προς Ασία όσον αφορά την επιρροή που θέλουν να ασκήσουν. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να βασιστεί τόσο πολύ στους Αμερικανού, πρέπει κινείται μόνη της. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε δικό μας δυναμικό στα κράτη-μέλη. Με προβληματίζει η ιδέα του, της άνωθεν επιβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέτρων. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων. θα επιβάλλουν οι δυνάμεις της αγοράς. Οι BA, οι ADS και οι μικρότερες εταιρείε θα πρέπει να ενοποιηθούν και αυτό θα συνεπάγεται διακυβερνητικά προβλήματα διασυνοριακά προς διευθέτηση. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτά που είπα, κυρίως όσον αφορά το Ελεύθερη συναλλαγή, ζώνη ελεύθερη συναλλαγό με, την, με τη ΣΥΠΑ. Και αν θα είναι εντός ή εκτός ε, της εντολής σας αυτή η συμφωνία στον τομέα. Ο κύριος Αγκουράκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα, θα είμαι από τους ε, λεγόμενους αφελείς από τον κύριο Επίτροπο ε, για τον εξής λόγο. Υπόθηκαν πολλά και καταλαβαίνω ότι έχετε και μεγάλες δυσκολίες κύριε Επίτροπε και τα πράγματα είναι απλά. Στην Ινδία από ό,τι γνωρίζω το Ραφάλ χτυπιέται με το Eurofighter ποιο από τα δύο θα πάρει η Ινδική κυβέρνηση η British Airspace, μαθαίνω, έφυγε από τις Ηνωμένε Πολιτείε για το cloud computing για λόγους φόβου ότι θα υπάρχει κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων από τους Αμερικανούς. Στην Ελλάδα η Ενίσα φεύγει από το Ηράκλειο, πάει στην Αθήνα, ενδεχομένως θα πάει και στη Χάγη. Είναι υπηρεσία για την προστασία ε, από τον κυβερνοπόλεμο, κύριε Επίτροπε. Ε, και αυτό διότι από ό,τι λέει μια μελέτη της Κομισιόν θα ενταχθούν όλα αυτά τα πράγματα στην ε, Europol. Στην Ελλάδα κύριε Επίτροπε, επειδή μιλήσατε για πολιτική και μη πολιτική έρευνα, θέλω να σας πω το εξής. Όπως αγνωρίζετε τα ελληνικά ναυπηγεία δεν μπορούν να κατασκευάσουν ε, μη πολεμικά πλοία αν δεν έχουν φυσικά κρατικές επιδοτήσεις. Μπορούν όμως κάλλιστα να κατασκευάζουν πολεμικά πλοία, ε, πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα οποία ως διαμαγείας είναι βεβαίως παραγγελίες ε, από γερμανικά ναυπηγεία. Το λέω αυτό κύριε Επίτροπε, διότι μας είπατε πάρα πολύ ωραία λόγια για την ε, αύξηση της αποδοτικότητας της έρευνας και για το δίθεν πρέπει να, να, να αποβάλουμε ιδεολογικά, όπως είπατε, όρια μεταξύ της στρατιωτικής και της μη στρατιωτικής έρευνας. Δεν είναι ιδεολογικά, κύριε Επίτροπε, τα προβλήματα. Είναι καθαρά πρακτικά προβλήματα. Στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, παραδείγματο χάρη, φαντάζουμε ότι σπουδάζουν φοιτητές και από άλλες χώρες. Από την Κίνα, από τη Ρωσία, δεν ξέρω από πού αλλού. Φανταζόσαστε εσείς σε Ιταλικό Πανεπιστήμιο να υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ στα οποία να έχουν πρόσβαση και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Αποκλείεται. Δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Φανταζόσαστε εσείς πανεπιστήμια σε αυτή την εποχή της κρίσης που υπάρχει να μην υπάρχουν πόροι κάποια πανεπιστήμια να θέλουν ε, μη στρατιωτική έρευνα όταν οι παχουλές, ε, πώς προσφορές θα είναι από την ε, πολεμική βιομηχανία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι θα τρέχουν σαν παλαδί να πάρουν στρατιωτικά προγράμματα. Τρίτο ζήτημα και σημαντικό, επειδή έγινε λόγος για συγχωνεύσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτά συμβαίνουν. Όμως, όπως γίνεται παντού, δημιουργούνται αυτά υποτίθεται για να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, Υποτίθεται για να μειωθεί το κόστος, αλλά στην πραγματικότητα ξέρετε τι γίνεται. Μονοπολείται η αγορά και αυτό που έχει το μονοπόλιο υπαγορεύει και τι τιμέ. Αυτό γίνεται παντού. Και το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην αμυντική βιομηχανία. Κλείνω κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι άλλα πράγματα είναι από πίσω. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια μεγάλη να γίνουν μεγαλύτερη και τελειώνω με το εξή απλό. Εάν πραγματικά και η Κομισιόν και ο, ο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ενδιαφερόταν να είναι πιο αποδοτική άμυνα, σας ρωτάω ευθαρσώς. Γιατί δεν ξεκινάει η συνεργασία από project που ξέρουμε ότι σας απασχολούν, αλλά δεν γίνονται. Παραδείγματος χάρη, δεν σας άκουσα να μιλάτε, για ένα ευρωπαϊκό μεταγωγικό μέσο ανεφοδιασμού στον αέρα, που δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν γίνεται λόγος γι' αυτό. Δεν σας άκουσα να μιλάτε για μία επανδρομένα πλοία. Δεν σας άκουσα να μιλάτε γι' αυτό. Δεν σας άκουσα να μιλάτε επίσης για το λεγόμενο pooling and sharing τελικά συνεργαζόσαστε με, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ή ο καθένα κάνει ό,τι νομίζει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ο κ. Σταγιάννη. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μου άρεσαν αυτά που είπε ο κ. Γιάννη σε αυτό το οποίο είπε. Και συμφωνώ βεβαίω μαζί του, λέει στα Ισπανικά ο Επίτροπο. Διότι νομίζω ότι κατάλαβε τι έργο επιτελούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, δεν θέλω να επιβάλλω αποφάσεις στα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ο συντονισμός της ε, βιομηχανικής πολιτικής, σύγχρονα της ε, πολιτικής που θα αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όχι, η Ευρώπη δεν είναι ΝΑΤΟ, είναι κάτι το άλλο. Και ξέρω είμαι παιδί του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί υπηρετούσε ο στρατηγικός ο πατέρας μου και φυσικά και δεν λέω ότι είμαι υπέρ κατά άλλο το ΝΑΤΟ, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάνει κάτι η Ευρώπη, το κάνει ως Ευρώπη. Αν το κάνει μια Ευρωπαϊκή χώρα, ως μέλος του ΝΑΤΟ, το κάνει το ΝΑΤΟ. Και όταν μιλούμε για την Ευρώπη, φυσικά και αυτό σημαίνει ότι είμαστε αντιαμερικανοί. Εγώ είμαι υπέρ της εμπορική συμφωνία με ΕΠΑ και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό για εμά να υπάρχει συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι είναι από τα, τους πιο σημαντικούς φίλους που έχει η Ευρώπη. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δουλεύω για την Ευρώπη. Δεν δουλεύω κατά του ΝΑΤΟ. Μπορώ, μπορώ το και το ένα να κάνω και το άλλο. ούτε το ότι υπηρετώ την Ευρώπη σημαίνει ότι είμαι κατά τον ΙΠΑ. Αν εγώ θέλω να ωφελήσω την οικογένειά μου, δεν σημαίνει ότι στρέφομαι κατά τη δική σου. Η οικογένεια τα Γιάννη, ένα πράγμα, και η, ε, οικογένεια Γιάννη είναι άλλο πράγμα. Επομένω, θέλουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, άμυνα. Ή θα προχωρήσουμε ή θα πεθάνουμε. Γι' αυτό και σα λέω ότι θα πρέπει να εκπονήσουμε μια πολιτική άμυνα για την Ευρώπη. Έχουμε εξωτερική πολιτική και χρειαζόμαστε και πολιτική άμυνας ευρωπαϊκή. Πώς να σταθεί η εξωτερική πολιτική, πώς να υπάρχει η πολιτική τη άμυνα. Ξέρω ότι δεν σα αρέσουν αυτά που λέει ο κύριε Τάνοκ, αλλά αυτή είναι η θέση που έχω. Democracy. We are in democracy. My position is not your position. Ε, τι να κάνουμε, δημοκρατία έχουμε λέει ο κύριος Επίτροπο. Άλλη δική μου θέση, άλλη δική σας. Είναι η προσωπική μου θέση. Ε, we are in democracy, freedom ε, also ε, Δημοκρατία έχουμε. Ελευθερία έχουμε. Και ακριβώ αυτό είναι το σημαντικό. υπάρχουν σε ένα διάλογο διαφορετικέ θέσει, διαφορετικέ ιδέε. Δεν ταυτίζει θέση με τη δική μου. Καλά. Ακριβώ το πιο σωστό είναι να μπορεί κανεί να τα Τέλο πάντων. Όσον αφορά τα άλλα θέματα δεν κατανόησα αυτά που είπε ο κ. Σαγκουράκης. Διότι κάποια πράγματα δεν είναι στην ανακοίνωση και δεν είναι στην αρμοδιότητα της ε, α, αμυντικής βιομηχανίας. Δεν μπορώ λοιπόν να παρουσιάσω πράγματα τα οποία δεν εμπεριέχονται στο κείμενο και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής. Βεβαίως, προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την ασφάλεια. Και το θέμα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε προτεραιότητες. Να έχουμε αντίσταση στον κυβερνοχώρο, να μειωθεί σημαντική εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Θέλουμε να εφαρμόσουμε πολιτική άμυνα στον κυβερνοχώρο σε σύνδεση με την πολιτική άμυνα και ασφαλεία στην κοινή, να αναπτύξουμε μηχανικού και τεχνολογικού πόρου όσον αφορά την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και να έχουμε διεθνή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κυβερνοχώρο και να προωθήσουμε την προστιθέμενη ασυξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της υπηρεσίας άμυνας για να αναπτυχθούν ε, για την προστασία των πολιτών μη επανδρομένα οχήματα, υπτάμενα οχήματα μάλλον εννοεί, τα drones. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις εκφράζω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μπορούμε πάντα να συζητούμε και αν υπάρχουν διαφορετικές ιδέες, αν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες μας, αν θέλουμε να έχουμε ε, καλές πολιτικές και στον τομέα της άμυνας, της αμυντικής βιομηχανίας των κρατών μελών, πιστεύω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, για τις διάφορες ε, κριτικές απόψεις που ακούστηκαν. Ε, είμαι έτοιμο να δεχτώ τυχόν έγγραφα που θέλουν οι Ευρωβουλευτέ να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν, παρουσιάσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Άμυνα για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε το διάλογο μαζί και ελπίζω να μπορέσω να σας παρουσιάσω το κείμενο μετά από την έγκριση του σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ένας που άνοιξε και θα συνεχιστεί. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόταση που κάνατε για να εμπλουτίσουμε ενδεχομένως τον προβληματισμό σας με τη συνεισφορά μας. Θα χαρούν πολύ ορισμένοι βουλευτές να στείλουν ε, προτάσεις ή αντιρρήσεις. Το λέω βλέποντας κάποιους συναδέλφους. Και μετά την ανακοίνωση, στο χρόνο μεταξύ ανακοινώσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι το Συμβούλιο, καλό θα ήταν ε, εδώ να έχουμε άλλη μια επαφή και με τον συνάδελφό σας, είσαι, τον ε, κύριο Μισελ Μπαρνιέ, να είσαστε και δύο παρόντες. Ε, και ταιριάζουν και αυτά που είπατε εσείς ε, με αυτά που μας είπε εδώ και μερικές εβδομάδες ο κ. Μπαρνιέ. Έχετε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ σας, ελευθερώνω. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι εσωτερικής αγοράς σας περιμένουν. Λοιπόν, γεια σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δοθεί της καθυστερήσεως. Καθίστε παρακαλώ λοιπόν για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με το Αφγανιστάν. Με τα χαράς υποδέχομαι δύο προσωπικότητες που ήδη συναντήσαμε και έχουμε εκτιμήσει τι ικανότητε του ο κ. Ουζάσκα, ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στο Αφγανιστάν μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά στη Μόσχα, στην αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω εκεί. Ήδη σα ακούσαμε αρκετέ φορέ, αλλά θα είναι ιδιαίτερο χρήσιμο να μα ενημερώσετε. Και ο στρατηγό Ντεμποβάνκοφ την προηγούμενη φορά που σα ακούσαμε, ήταν σε βιντεοδιά... βιντεοδιάσκεψη από την Καμπούλ σας ευχαριστούμε, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Μετά το Στρασβούργο βέβαια, διότι είσαστε στο Καμπούλ σαν επικεφαλής του επιτελείου της Ιουσάφ, αλλά πάντα ήσασταν διοικητής του Eurocore. Καταφθάνετε στην ώρα σας από το Στρασβούργο. Άρα λειτουργούν ε, οι διασυνδέσεις. Στην ΙΣΑΦ είσαστε πάνω από ένα χρόνο στην Καμπούλ επικεφαλής και θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως να ξέρουμε τι μαθήματα αντλείται όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, όσον αφορά την ασφάλεια και το μέλλον που είναι γεμάτο αβεβαιότητα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ χθες συνεδρίαζαν και σήμερα στις Βρυξέλλες για να δουν τι συνέχεια θα δοθεί, τι θα ακολουθήσει μετά το 2014 στο Αφγανιστάν, Μεγάλη αβεβαιότητα και ερωτηματικά απομένουν όσον αφορά τις δυνάμεις που θα παραμείνουν, την εντολή που θα έχουν, τη χρηματοδότηση των αποστολών που θα παραμείνουν. Δεν περιμένουμε απαραίτητα σήμερα πως σας απαντήσει αυτά, αλλά θέλουμε μία ενημέρωση. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας μετά τη μακρά διαμονή σας εκεί, τι μπορούμε να περιμένουμε και τι μπορεί να γίνει για να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η ευαίσθητη μετάβαση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που είμαι ανάμεσά σας σήμερα το απόγευμα για να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά το Αφγανιστάν, λέει ο κ. Ζάσκας. Ο φίλος μου, ο στρατηγός Δεμπαβίνκοφ ε, χαίρομαι που είναι εδώ μαζί μας για τη συζήτηση. Κυρίε και κύριοι, με τα χαρά σε επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες για τι εξελίξει στο Αφγανιστάν, κυρίως όσον αφορά τη μετάβαση, μελλοντικέ προοπτικές και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο Αφγανιστάν πριν και μετά το 2014. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής τα τελευταία 10 χρόνια έχουν ε, αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν για να μην γίνει ασφαλής ε, περιοχή για του τρομοκράτε που απειλούν τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα για να μειωθεί η φτώχεια, αυτή η προσπάθεια και να βελτιωθεί ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να βελτιωθεί η δημοκρατία. Υποστηρίζουμε το Αφγανιστάν μέσω ολιστική προσεγγίσεω που εξασφαλίζει συμπράξει μεταξύ πολιτικού τομέα, τομέα ασφάλεια και των διαφόρων προσπαθειών Προσπαθούμε να υποστηρίξουν την καλή διακυβέρνηση, να μεταρρυθμιστεί ο δικαστικό τομέα και να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα πιστό και ισχυρό εταίρο του ΟΗΕ και των αποστολών στο Αφγανιστάν και εκπληρεί την εντολή που έχει ανατεθεί για την προετοιμασία για τι εκλογέ, κυρίω ενώ πλησιάζουν οι προεδρικέ εκλογέ τον Απρίλιο του 2014. Μέσω του UPOL συμβάλαμε στην αυξάνιση τη εθνική αστυνομία να γίνει επαγγελματική αστυνομία ικανή και με αναπτυξιακά μέσα συμβάλαμε τα μάλα όσον αφορά την υγεία και το γεωρικό τομέα. Και τα κράτη-μέλη αυτή είναι στο Αφγανιστάν για μακρό χρονικό διάστημα. Έχουμε αναλάβει υποχρεώσει να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και το λαό πολύ μετά το 2014. Η Αφγανική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει και άλλα βήματα εφαρμόζοντα αναγκαίε μεταρρυθμίσει για την ορθή διακυβέρνηση, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτω ώστε εμεί να μπορούμε να εκπληρώσουμε τι δικέ μα υποχρεώσει. Είναι προφανή τα κέρδη από τη μετάβαση αλλά είναι εύθραυστα τα κέρδη αυτά και μπορούν να έχουμε επιτυχία μόνο αν τα αποτελέσματα αυτά εδράζονται τη ορθή διακυβερνήσεω. Αν θέλουμε να είναι ε, ε ασφαλή η μετάβαση, πρέπει να κινηθεί πολιτικά. Ο στρατό υποχωρεί και δίνει το χώρο του στον πολιτικό κόσμο. Λοιπόν, Έχουμε, λάβει, έχουμε συνεργασία με τι δυνάμει ασφαλεία στο Αφγανιστάν και δώσαμε και τη σωστή υποστήριξη για να βοηθήσουμε. Οι κατασκευέ και η οικοδόμηση και οι μεταφορέ είναι κάτι δύσκολο λόγω ελλείψεω υποδομών και διότι δεν έχει μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη επιρροή η κεντρική κυβέρνηση. Δεν φτάνει μακριά. Έχουμε θετικέ εξελίξει, πρέπει να τι παραδεχτούμε. Το Αφγανιστάν έχει πετύχει την τελευταία δεκαετία ορατέ πρόοδου. 65% του πληθυσμού τώρα έχει πρόσβαση σε βασική περίθαλψη. Το 2002 ήταν 9%. Ελήφθησαν μέτρα για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και να υπάρξει πρόσβαση στην παιδεία. Δύσκολο. Το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν, είχε τα χάλια του μετά από δεκαετίες μαχών και επιθέσεων από πλευρά τη κυβέρνηση Ταλιμπάν κατά του εκπαιδευτικού συστήματο. Το 2002 λιγότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά ε, ήταν στην ε, επίσημη παιδεία, είχαν ε, εγγραφεί. Τώρα έχουν πάνω από 6 εκατομμύρια παιδιά έχουν εγγραφεί. Υψηλότερος αριθμός στην ιστορία του Αφγανιστάν. 2,7 εκατομμύρια κορίτσια. Το Αφγανιστάν έχει τεράστιο δυναμικό για οικονομική ανάπτυξη. Και αναπτύσσεται η οικονομία τα τελευταία χρόνια 9 με 11% το χρόνο. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με τη σταδιακή απόσυρση της διεθνούς υποστήριξης αυτή η ανάπτυξη θα μειωθεί. Επιπλέον, 8.000 χιλιόμετρα εθνικών αυτοκινητόδρομων, περιφερειακών δρόμων ε, έχουν κατασκευαστεί και μειώθηκε ο χρόνος ταξιδίων κατά 75% μεταξύ διαφορών κέντρων. Η πρόσβαση στον ηλεκτρισμό αυξήθηκε κατά 250%. Πάνω από 30% του πληθυσμού έχει ηλεκτροδότηση διεθνής εκπαίδευση εστιάζεται στην εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν σε θέματα μιλητίας διοίκησης, ιατρικής περίθαλψης και δημιουργίας ειδικών δυνάμεων. Όμως, η ΙΝΑΣΕΦ ε, δεν, έχει, δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορεί να αναλάβει ε, πλήρω την ασφάλεια. Ο στρατηγό Καρύμ έκανε σαν επικεφαλής του επιτελείου είπε ότι μόνο μερικές μεραρχίες από το σύνολο μπορούν να επιχειρούν ανεξάρτητα. Εν γέννη. Οι διάφοροι ηγέτες, ε, οι οπλαρχηγοί, οι τοπικοί έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Κυρίως εν ώψη των εκλογών βλέπουμε να αλλάζει το τοπίο το πολιτικό στη χώρα. Νέες συμμαχίες, νέα πολιτικό κόμματα. Όμως με τη συμμετοχή παλαιών πολέμαρχων παίζουν βασικό ρόλο. Το 2015 το Αφγανιστάν πιθανότατα θα είχε, θα είχε ασφάλεια πολυεπίπεδη, θα ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και επιρροή τη κυβέρνησης θα ποικίλει. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική αστυνόμευση ε, και να παίρνει τη θέση των παραστατικών δυνάμεων. Πρέπει να υπάρξει επαγγελματική αστυνόμευση της χώρας. Υπάρχει και ένας κίνδυνος όλα όσα πετύχαμε σε 10 χρόνια, με έντονε προσπάθειε για δημιουργία θεσμών και για ανάπτυξη, όλα αυτά σταδιακά να καταρρεύσουν μετά το 2014. Όμω, δεν είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο. Αν εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Περιφερειακή φορεί και η διεθνή κοινότητα προωθήσουμε ένα συνέστημα εμπιστοσύνη και ιδιοκτησία, να θαρρυνθούν οι Αυγανοί και η Αυγανική κυβέρνηση, και αν η βιανική κυβέρνηση τηρήσει υποσχέσει τη. Αν γίνουν όλα αυτά, πιθανότατα θα έχουμε αργή αλλά σταθερή πρόοδο. Θα γίνεται πιο δημοκρατική η χώρα και πιο σταθερή. Αυτή η πρόοδο σίγουρα θα κλονιστεί από διάφορα προβλήματα και κρίσεις. Αλλά δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε το μέλλον ζωφερό. Η διεθνής κοινότητα θέλει να στηρίξει το Αφγανιστάν και πέρα το 2014. Το είδαμε από διάφορε στρατηγικέ συνεργασίε και σχετικέ συμφωνίε που υπεγράφησαν από πολλέ χώρε. Και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση τελειώνει τι διαπραγματεύσει για δεκαετή συμφωνία συνεργασία για σύμπραξη και ανάπτυξη με το Αφγανιστάν. Το Σικάγο και το Τόκιο ε, οδήγησαν σε δεσμεύσει των ερήφθη εναντίον του Αφγανιστάν για την υποστήριξη των εθνικών ε, δυνάμεων του Αφγανιστάν. Μεγαλύτερη πρόκληση είναι η χρηματοδότηση για τι εθνικέ δυνάμει ασφαλεία του Αφγανιστάν. Στο Τόκιο πέρσι η διεθνή κοινότητα δεσμεύτηκε να δώσει πάνω από 16 δις δολάρια, είπα, για μια τετραετία και να συνεχίσει την υποστήριξη μέχρι το 2017. Στα επίπεδα της περασμένης δεκαετίας, για να εξασφαλίζεται η συνεχής οικονομική ανάπτυξη και να μεταμορφωθεί το Αφγανιστάν. Χρειάζεται αυτό. Για να μπορεί να έχει χρήματα η κυβέρνηση του Αφγανιστάν πριν αρχίσει να έχει εισοδήματα δικά της. Και να μπορεί να γίνει αυτάρκη. Για πρώτη φορά αυτέ οι διεθνεί υποχρεώσει δίδονται προϋποθέσεις. Εξαρτώνται από την προθυμία να ανταποκριθεί και το Αφγανιστάν τι δεσμεύσει που ανέλαβε στο Τόκιο. Διαφανεί αξιόπιστες εκλογέ του 2014 με θεμητό αποτέλεσμα, υποστήριξη κατά πόση διαφθοράς, η πρόθεση τη δικαιοσύνη, βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίω των γυναικών, υποστήριξη οικονομική ανάπτυξη και να υπάρχει καλύτερη διαχείριση ε, του δημόσιου τομέα, κυρίως στο τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα της μεταρρύθμισης που συμφωνήθηκε στο Τόκιο και στο Σικάγο ε, είναι κάτι πολύ φιλόδοξο πράγματι και η εφαρμογή ε, απεδείχθη δύσκολη και αργή. Πολιτικά ζητήματα συνδυάστηκαν με προσδοκίες, δηλαδή ότι θα εξακολουθήσει η χρηματική ροή. Τώρα μας πρέπει να δεχθούμε ότι οι Αφγανοί θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτές οι αμοιβέ δεσμεύσει ε, δίδονται, έχουν αληφθεί υπό όρους για να υπάρξει αξιοπιστία, διατηρηθεί αξιοπιστία. Είναι σημαντικό λοιπόν, τώρα που σας μιλώ, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, τα, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να ξέρουν τι προσπάθειε κάνουμε στο Αφγανιστάν. Είμαστε υπόλογοι στου φορολογούμενου εμεί, στι πατρίδες μα. Πέρσι, στο δικαστικό τομέα, στη μεταρρύθμιση είχαμε ελλείψει και εμεί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πήραμε απόφαση να καθυστερήσουμε την ε, υλοποίηση της υποχρεώσεως για 20 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον τομέα μέχρι ότου να υπάρξει μια συμπεφωνημένη συγκεκριμένη στρατηγική στον τομέα αυτό. Εξάλλου, αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο ως μέλος της ομάδας 5 συν 3, που είμαστε δωρητές δηλαδή στην ε, παρακολούθηση των υποχρεώσεων που έχουν αληθεί στο Τόκιο και από τον Ιούλιο του 2013. Εν τέλει, όμω, η αφγανική κυβέρνηση θα χρειαστεί να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τι ευκαιρίε αυτέ και να δημιουργήσει βιώσιμο μέλλον για τον αφγανικό λαό. Οι Αφγανοί πρέπει να καταλήξουν ωστόσο σε ενότητα και συνοχή και συνεργασία μεταξύ των θεσμών του. Δεν θα πρέπει να αναμένουμε θαύματα ή κάποιε εμβαλωματικέ λύσει στην ε, χρονιά που μένει ακόμα τη ε, διακυβέρνηση Καρζάη. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι Αφγανοί πολιτικοί ηγέτες να αναλάβουν τα ενία της διακυβέρνησης, καθώς πλησιάζει το 2014. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνολό τους, την διασφάλιση της δημοκρατίας και τη δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά μέχρι τώρα έχουν βασιστεί στις δωρεές των δωρητών, στις διεθνείς δωρεές. Οποιαδήποτε λοιπόν ε, πρόοδος κινδυνεύει να απολεστεί η καθυστέρηση στον διορισμό των Αφγανών επιτρόπων, ήδη 1,5 χρόνο δηλαδή, θεωρείται ως ένα παράδειγμα της έλλειψης δέσμευσης της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Και όπως γνωρίζουμε, το πρόβλημα της αφγανικής ασφάλειας δεν μπορεί να λυθεί χωρίς συμμετοχή των τοπικών παραγόντων. Χρειάζεται και έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Η διαδικασία Heart of Asia ξεκίνησε στην Ιστανμπούλ το Νοέμβριο του 2011 για να προωθήσει τη σταθερότητα, ακαιρεότητα και ευημερία του Αφγανιστάν μέσα από μια σειρά μέτρων αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Πέρα, πέρα από αυτό, ως Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουμε ότι η ειρήνη στο Αφγανιστάν θα πρέπει να βασιστεί σε μια πολιτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς, stakeholder. Έχουν γίνει βήματα σε διάφορα επίπεδα, αλλά ακόμα συγκεκριμένες εξελίξεις είναι πολύ περιορισμένες. Ως παράδειγμα της συμφιλίωσης και της περιφερειακής συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στην υποστήριξη πολιτικά και οικονομικά της ικανότητας της αφγανικής κυβέρνησης να συμβάλλει στο διάλογο στην περιφέρεια, έτσι, στην περιοχή αυτή δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει νέα ε, συνεργασία και διασύνδεση. Και βεβαίως να μπορεί να ελέγχει τα σύνορά τη. και να ε, διοικεί τα τελωνία της. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Και το Αφγανιστάν και το Πακιστάν έχουν δείξει ότι αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο το πόσο αλληλοεξαρτώνται και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την σύγκρουση και τον ε, ε, φανατισμό στη ρίζα του. Είναι μακρά η διαδικασία για την συμφιλίωση αυτή και πρέπει να βασίζεται σε μια βάση ρεαλισμού. Είναι σημαντικό και οι χώρες αυτές να πάψουν να κατηγορούν η μία την άλλη δημοσίως. Η συμφιλίωση του Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι μια διαδικασία η οποία θα κυριαρχείται από τους ίδιους τους Αφγανούς. Και βεβαίως και με σεβασμό του αφγανικού συστήματος και των όσων προβλέπει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίω για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι χώρες μέλη έχουν συμβάλει σε θετικές πρωτοβουλίες για να υποστηρίξουν αυτό τον ενδοαφγανικό διάλογο με την πρωτοβουλία Σαντιγή καθώς και με τριμερείς ε, ε, επαφές της ΕΕ. Βασιζόμενοι στη μακρά μας εμπειρία διαχείρισης κρίσεων εκπαιδεύουμε την Αφγανική Εθνική Αστυνομία με την ε, αποστολή CSTP, την EUPOL, καθώς και άλλους οργανισμούς, ΛΟΤΦΑ κλπ. Στις επικείμενες εκλογές που θα είναι κρίσιμες για την περαιτέρω πορεία του Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την UNDP Elect 2, όχι μόνο τεχνικά, για να διεξαχθούν σωστά οι εκλογές, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η διεξαγωγή των εκλογών, εκλογών θα γίνει με τρόπο που να περιλάβει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως βασικός δωρητής της ΕΛΕΚΤ 2, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει με 10 εκατομμύρια ευρώ στο Instrument for Stability για να υπάρξουν πιο διαφανείς θεσμοί οι οποίοι θα προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον αφγανικό λαό. Εμείς υποστηρίζουμε το Αφγάνιστάν στη δημόσια διοίκηση και στην υγεία. Ένα οριζόντιο θέμα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, γιατί η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Με συνολική αντιμετώπιση όλου του προβλήματος και από άψη υγείας και από άψη ελέγχου συνόρων κλπ. Τέλος, εμείς ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών να πάυσουν την βία κατά των γυναικών, να σταματήσουν τους αναγκαστικούς γάμους και να προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο στις γυναίκες που έχουν ανάγκη. Κυρίε και κύριοι, ως επικεφαλής της αποστολής στο Αφγανιστάν εδώ και τρία χρόνια, έχω διαπιστώσει την ε, πρόοδο που έχουμε επιτελέσει συλλογικά στο Αφγανιστάν. Μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει το 2014, όμως οι ρίζες της σύγκρουσης, ο φανατισμός, ο αναλφαβητισμός, η φτώχεια, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν. Όλοι πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να επαναλάβουμε τα σφάλματα του 1989 ή το 2002. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Αφγανιστάν σε όλη αυτή τη δεκαετία μεταρρύθμισης. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα μέσα. Να στηρίξουμε και τους γείτονές του. Οι Αφγανοί μας εταίροι πρέπει να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους πολύ πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Η υποστήριξη που υποσχεθήκαμε στο Σικάγο και στο Τόκιο θα συνεχιστούν μόνο εάν οι προεδρικές εκλογές του 2014 γίνουν με τρόπο που να μην αποκλείει κανένα και να είναι δημοκρατικός και να γίνουν γνήσια βήματα για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών και να υπάρξει κλίμα για οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό τον ευρύ διάλογο θα πρέπει εμείς να παίξουμε επικοδομητικό ρόλο. Εάν απογοητευτούμε από την έλλειψη απόδοσης θα μειωθούν οι προσπάθειες. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η σταθερότητα που έχει επιτευχθεί με τόσο υψηλό τίμημα, θα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση των εθνικών αφγανικών αρχών. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν είναι μακροπρόθεσμη. και αναμένουμε την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν για φέτος ήδη. Βασισμένη στην ιστορική μας εμπειρία θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να εμπνέουμε την συμφιλίωση. Να ρίξουμε το βάρος μας στην ενίσχυση του capacity building, το κράτος δικαίου, την ε, δημιουργία και εκπαίδευση μη στρατιωτικής αστυνομίας, civilian police και αυτά να γίνουν με χρήση κάθε δυνατής ευκαιρίας, κάθε, δυνατή, κάθε δυνατότητας για συλλογική χρήση όλων των πόρων ώστε να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο Αφγανιστάν τον χρόνο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να καθορίζουμε προτεραιότητες και να ενισχύουμε την υποστήριξη στο Αφγανιστάν σε αυτή την δεκαετία της μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, ειδική επιστολμένα. Δεν πάμε ότι αυτό αποτελεί απολογισμό όταν έχετε κάνει διαιτητή τη αποστολή σα, γιατί ακόμη χτυπώντας μπροστά σα. Τέλο πάντων, πρόκειται για μια σφαιρική προσέγγιση για όσα έχουν γίνει και ευχαριστούμε για την τόσο πλήρη έκθεση πεπραγμένα που μα κάνατε. Στρατηγία μου τώρα, για πετε μας ε, από πλευρά ασφαλείας, ε, εσείς θα μας τα πείτε, φαντάζομαι. Είστε και επικεφαλής της ΕΣΑΦ πάνω από ένα χρόνο. Έχετε την σκητάλη. Κατόπιν τον όσων είπε ο κύριο Πρέσβης, ο κύριος Ουσάσκας, να μην επαναλάβω τα ίδια βεβαίω και συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπε, με το τοπίο που μας το περιέγραψε, ε, μας τα είπε με τρόπο ταυτοχρόνως ε, ρεαλιστικό το Αφγανιστάν και ταυτόχρονα λέω θα πρέπει να επιδείξουμε στάση υπομονής για να αποκτήσει ανάπτυξη η χώρα όπως είναι οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες μας. Στα λεπτά που μου αναλογούν να σας πω δύο λόγια και μετά να απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις να σας απαντήσω υπό πολλές ιδιότητες που έχω σε αυτή την αποστολή των 15 μηνών στο πλάι του στρατηγού Αλέν, επικεφαλής του επιτελείου του, σε συνεργασία με τις Αμερικανικές Δυνάμεις και, στο, και του ΝΑΤΟ. Έχουν περίπου εκεί 150.000 άνδρες, εκ των οποίων 100.000 είναι Αμερικανοί επίσης. Και ότι αυτή η ρόλη λοιπόν που διαδραμάτισα δεν είναι αντιφατική. Ε, είμαι διοικητή των γαλλικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Και αναπτύχθηκε στην Καμπούλ το ε, σώμα των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και με βάση το Στρασβούργο ξεκινήσαμε και διαρθρώθηκε έτσι η σάφη στις διαφορετικές της ε, πτυχές. Όσον αφορά το, το Αφγανιστάν, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύνοψη των όσων διαπιστώνουν ότι ισχύουν για αυτή τη χώρα, θα μπορούσα να πω ότι όλοι είχαμε πάρα πολύ βάλει ψηλά τον πύχη όταν είπαμε ότι στόχος μας είναι αυτός που είπαμε, χωρίς όμως χωρίς να λάβουμε υπόψη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα το 2001, στην αρχή δηλαδή της διαδρομής. Δεν είχε σύνταγμα. Δεν είχε θεσμικά όργανα. Δεν υπήρχε δικαιοσύνη. Δεν υπήρχε κεντρική η κυβέρνηση, περιφερειακές ε, αρχές. Δεν υπήρχαν ε, διοκτικές αρχές, δυνάμεις ασφαλείας, οργάνωση κρατική, ε, ήταν μέσα σε βαθιά φτώχεια η χώρα και ακόμα είναι μια χώρα όπου κυριαρχεί η καλλιέργεια το, για το πόρο των εργοτικών όπως το 95% το οποίο προέρχεται από το Αφγανιστάν. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε υπό καλύτερου όρου και θα μπορούσαμε την επόμενη φορά να πούμε ότι ε, θα θέλαμε τα πράγματα να είναι απλούστερα για να υλοποιήσουμε αυτό το οποία θέλουμε. Και εδώ και αρκετό καιρό ακούμε κάποιες ε, επικρίσεις κυρίως από αμερικανικής πλευράς αλλά και ευρωπαϊκής από Βρετανία, από Γαλλία και υπάρχουν επικρίσεις σε σχέση με τα λάθη τα οποία διαπράξαμε στο Αφγανιστάν. Βάσει αυτής της κριτικής υπάρχει τα ακούω αυτά, αλλά τα φιλτράρω από πλευρά του ότι εγώ δρώ εκεί, επί τόπου. Πάντω, αυτό το οποίο όλοι θα πρέπει να πούμε είναι ότι, ότι πρόκειται για ένα συνασπισμό, για μια συμμαχία 50 χωρών που δρούν στο Αφγανιστάν. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε και αυτό που πραγματικά έπρεπε να, να, να, να πούνε να μα επικρίνουν ότι δεν καταλάβαμε σε ποια κατάσταση ε, βρίσκεται η χώρα μετά από 30 χρόνια εμφυλίου πολέμου και πολέμου. Και με ένα τέτοιο καθεστώς το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Επομένω, έτσι προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας. Καλά, εγώ ε, ήρθα στην τελευταία φάση αυτής της διαδρομής, αλλά βέβαια τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική η φάση αυτή, γιατί ο χρόνος δουλεύει εναντίον μας. Και δεν μπορούμε παρά να είμαστε περήφανοι για όσους έχουμε επιτελέσει. Γιατί για το ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει σταθερότητα ούτε το 2014, ούτε το 2025 από πλευρά ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Ίσως το 2060, το 2070 να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ο προηγούμενος ε, πρέσβης, ο αντίστοιχος του Τζον Άλεν, ήταν ε, ε, Βρετανός, είχε διατελέσει πρέσβης στο Ιράν. Ήταν ο ειδικό απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέως του ΝΑΤΟ. Αποχωρώντας, είπε μερικά πράγματα που τα κρίνω πάρα πολύ εύστοχα. Και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί με τον κ. Μέσα σε 40 χρόνια θα δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας. Επομένως, υπομονή. Αλλά Ποια είναι η δυσκολία. Εμείς όλοι που προχώμαστε από ανεπιγμένες χώρες, συνήθως δεν έχουμε αυτή την αρετή της υπομονής. Είμαστε ανυπόμονοι. Επιζητούμε αποτελέσματα, αποτελέσματα τα οποία να τρέφουν και τροφοδοτούν τα ΜΜΕ και την πολιτική. Όμως αυτή η ανυπομονησία δεν έχει καμία σχέση με την αντίληψη της πολιτικής του, του, και του χρόνου ή στο Αφγανιστάν, που εκεί ο χρόνος, με τη δική του αντίληψη, περνάει πολύ πιο αργά από ό,τι για μας εδώ. Επομένως, δεν κάναμε τη σωστή εκτίμηση των πραγμάτων. Όπως σας είπα, ή επίσης την απουσία της παιδεία, γιατί όλα, όλα, όλα τελικά έχουν να κάνουν με την παιδεία. Και η παιδεία, η κατάσταση παιδείας στη χώρα εκείνη, Τώρα... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνει κάποια αισιοδοξία, αλλά όχι τόσο πολύ. Γι' αυτό το λόγο θα λέω και εγώ γαλλικά και όχι αγγλικά, γιατί είναι αλήθεια. ξέρω ότι τα, τα στοιχεία δεν είναι τόσο αισιόδοξα, αλλά έχουμε, είπαμε, 9 εκατομμύρια παιδιών ε, που πάνε τώρα στο σχολείο ε, περισσότερο από το 2005 και 8 εκατομμύρια είναι τα ε, κορίτσια και τα αγόρια και έχουμε είπαμε 70% των ανηλίκων οι οποίοι φοιτούν σε σχολείο. Άρα 30% δεν πάνε στο σχολείο. αυτό που να πει αυτή στατιστική. 30% των ανηλίκων είναι αγράμματοι. Δεν πάνε στο σχολείο. Δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στη γνώση, στην παιδεία και 40-50 χρόνια εκεί θα, θα, ζουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι και στη χώρα. Άρα η προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει για την παιδεία στο Αφγανιστάν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τουλάχιστον έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου και για αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κάνει βήματα προόδου γενικότερα η χώρα. Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ε, δηλαδή ήταν εκεί πέρα πρωτοπόροι. Ε, κατασκευάσαμε 450 σχολεία και επικεντρώντας προσοχή μας δηλαδή στην παιδεία θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε μία ή δύο γενναίες τα παιδιά που πήγαν στο σχολείο 2005-2006 θα είναι στα πράγματα του 2040-2050. Πολλές φορές πολλά think tank αντιμετωπίζουν το Αφγανιστάν όπως το λέγαμε παλιά, όπως το βλέπαμε παλιά, δηλαδή Τατζίκι και Παστούν. Όμως υπάρχουν ακόμα δυσκολίες, λέμε. Και θα υπάρχουν δυσκολίες για τη χώρα και στο μέλλον. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο που θα έχει η χώρα είναι η σύγκρουση των γενεών. Οι παλιοί από τη μια, οι πολέμαρχοι, οι οποίοι και σήμερα είναι στα πράγματα ως επιτοπλίστων. και από λάς κεντρικής κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών. Αυτοί, περισσότεροι από αυτούς, δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, είναι αγράμματοι. Αλλά από την άλλη μεριά είναι η νέα γενεά, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της πρόσβασης στην παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, τα οποία διαθέτουν τα σύγχρονα, και αυτοί όλοι θα έχουν άλλες μεθόδους, μέσα, όραμα για το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Τελείως διαφορετικά από ό,τι οι παλιότεροι. Θα γίνει λοιπόν σε αυτή η σύγκρουση των γενιών 2025, 2030, 2035. Αναπόφευκτα θα γίνει διαφορετική κατανομή της εξουσίας σε σχέση με το σήμερα. Κάτι άλλο, το τέταρτο, η ουσία του ζητήματος. Όλοι σε επίπεδο στρατιωτικό, βέβαια, ενώ την διεύθυνση και με μεγάλη ικανότητα την ε, είχαν οι Αμερικανοί, κάνουν μεγάλο λάθος. Όταν έχουμε εξέγερση, αυτή τα πλασματικά μόνο, μόνο από τους ντόπιου. Δεν γίνεται καταστολή από ξένους. Οπότε και εκεί κάναμε λάθος και χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Φτιάξαμε τον Εθνικό Αφγανικό Στρατό από το 2007-2008 και μετά από είπε ο κύριο Πρέσβη. Θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει την πρώτη ενδεκάτου του 2001. Οπότε και στατορίσαμε περίπου 350.000 δυνάμεις ασφαλείας. Ντόπιου από την αστυνομία ή από το στρατό. Και προσπαθήσαμε να στατολογήσουμε τους καλύτερους και να ετοιμάσουμε κάποιες ειδικέ δυνάμεις οι οποίες σήμερα δραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ειδικέ δυνάμεις που είναι πολύ αποτελεσματικοί για την ε, αντιμετώπιση των πιο σκληρών από τους αντιπάλους μας εκεί. Επίσης, στρατολογήσαμε με ένα αμερικανικό πρόγραμμα αυτό που είπαμε αφγανική τοπική αστυνομία. 30.000 τοπικοί αστυνομικοί προσελήφθησαν οι οποίοι με την παρουσία τους κατόπιν εκπαίδευσης εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Ήταν 30.000, σήμερα είναι περίπου 22-25 και θα φτάσουν τους 45.000 το 2015-16. Και έχουμε επίσης και κάποιους σεκιουριτάδες, 22.000 αυτή είναι οργανωμένη από τον, κάποιο τρόπο σαν ιδιωτικό φορέα και ε, αυτοί οι φυλάσσουν ε, πράγματι περιουσία κυρίω. Οπότε το σύνολο όλων αυτών 2014-2015 θα είναι περισσότερο από 400.000 είναι όλοι οι οποίοι βιαστικά επιστρατεύτηκαν, πολύ βιαστικά εκπαιδεύτηκαν, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτοί δεν αποτελούν μια εθνική δύναμη η οποία θα δώσει τη μάχη της και με επιτυχία, γιατί το έκαναν αυτό. Είναι αποφασισμένοι για δράση. Βεβαίω υπάρχουν κάποια προβλήματα, Υπάρχουν ε, προβλήματα οργάνωσης, ε, ηγεσία, συντήρησης του υλικού των οχημάτων, οικονομικά, ε, καύσιμα. Δεν, λέμε ότι όλα είναι τέλεια και ιδανικά. Όμως, δεν μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο έχει λεχθεί πρόσφατα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν θα καταρρεύσουν άπαξ και οι ξένοι φύγουν. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Ούτε ένα το δεν πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο. Δυσκολίε θα υπάρξουν, αλλά να καταρρεύσουν, όχι. Εκτό αν θεωρήσουμε ότι όλε αυτέ τι προσπάθειε που σα είπα θα ε, σταματήσουν. Θα σταματήσουν πριν περάσει η δεκαετία που σα είπα. Οι προσπάθειε αυτέ σε σχέση με τι δυνάμει ασφαλεία και σχέση με το κράτο στο Αφγανιστάν. Τώρα, τελευταίο σημείο που θέλω να σας αναπτύξω είναι οι δυνάμεις της συμμαχίας. Πριν από αυτήν εδώ τη συζήτηση είχε προηγηθεί κάποια άλλη όπου είχαμε ε, αναπτύξει την ιδέα ότι οι Αμερικανοί μας σύμμαχοι πώς συντονίζονται με τις δικές μας ε, δυνάμεις τις ευρωπαϊκές. Εγώ έχω τρεις ρόλους. Ως ε, Γάλλος, ως ε, αξιωματικός του, του, ΝΑΤΟ και επίσης ως Ευρωπαίος, ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Στατιωτικού Σώματος. Κανένα πρόβλημα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, όσον αφορά τη χάραξη στρατηγικής, την χρήση του υλικού, όσον αφορά τον καθημερινό ε, διάλογο ή όποτε γίνεται τέλο πάντων με τους πρέσβεις του και τα ξέρει ο κύριος Σάσκας. Πολλές φορές συναντώμεθα ε, φιλικά ή και επαγγελματικά, αλλά τόσο αυτό ισχύει για όλους τους πρέσβεις που παρίστανται στην Καμπούλ, το, τον Βρετανό πρέσβη, το, το Γάλλο, τον Αμερικανό. Συγγνώμη, ξέχασα κάποια χώρα γιατί συνεργαζόμαστε. Ε, υπάρχει κατανόηση και επιζητούμε να ακούγεται ενία η φωνή μας, προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης, πώς θα βοηθήσουμε τους Αφγανούς. Δεν είμαστε εκεί για κάποιο δική μας φιλοδοξία. Προσπαθούμε να έχει αυτή η χώρα ένα μέλλον καλύτερο το παρελθόν των τελευταίων 30 ετών. Οπότε γι' αυτό στρεφόμεθα προς τους ε, Αφγανούς και τους λέμε ότι θα πρέπει αυτοί να δουν και να επισημάνουν τι χρειάζεται, τι χρειάζονται. Και εκεί είναι η δυσκολία. Και είναι δυσκολία που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. ότι δεν είχαμε ως συνομιλητή μία κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που να είναι αυτό που εννοούμε εμείς κυβέρνηση. Δεν είχαμε απέναντί μας μία ε, διοίκηση που η λήψη να μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Είναι κάποιο δίκτυο κοιτικό τέλο πάντων που ας πούμε στην επαρχία του Χέλμαντ να, να μπορεί να δράσει να υπάρχει εκεί. Αυτή ήταν ακριβώς η δυσκολία. Αυτή η τελευταία μου επίσκεψη, να σας πω έτσι ε, ενδεικτικά, η τελευταία μου επομένως ε, επίσκεψη επιτόπου ήταν μέσα Ιανουαρίου φέτος. Και και εκεί είχα τον Ρίτσαρτ Σέφερ και πήγαμε στο Χέλμοντ. Αυτό είναι ε, ε, ε, στρατηγός Άγγλος. Πήγαμε εκεί, είδαμε έναν υποδιοικητή, υποκυβερνήτη, αν, αντικυβερνήτη, αυτός ο οποίος ε, είχε διοριστεί, ε, ήρθε από την Καμπούλ, είχε πάει σε πανεπιστήμιο, ήταν νέο δυναμικό. Κά, κάτι περίπου σαν υπο υποπεριφερειάρχη στην, ε, στη Γαλλία και ασχολείται με ασφάλεια, με παιδεία, με, με, με, το υδροδότης, τόσο ε, ό,τι περιφερειακές ειδικέ αρμοδιότητες υπάρχουν. Και εγώ με, και, ο Ρίτσαρτ λοιπόν, ο συνάδελφος, συζητήσαμε με αυτόν και μετά φάμε, είπαμε, ρωτήσαμε πώς, πώς, πώς λειτουργεί εδώ το σύστημα. Αυτός μας είπε ότι μόνος του ήταν, μόνο εκείνος υπήρχε. Δεν είχε άλλο προσωπικό υποβοηθητικό. Αυτά στο Χέλμαντ, αλλά θα μπορούσαν να ισχύουν και άλλου στη χώρα. Ήξερε όμω αυτό τι προβλήματα είχε όσον αφορά την περιοχή του. Όμως δεν πτωήθηκε ήθελε να φτιάξει δρόμους, να φτιάξει σχολεία, ήταν αποφασισμένος να βελτιώσει την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση και ήξερε ότι μπορεί κάτι να κάνει όσον αφορά την ασφάλεια και ότι επίσης ο ρόλος ήταν πολύ σημαντικό για τον συντονισμό του δυνάμεων ασφαλείας. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω. Διότι αυτό θα να πω εγκατακλείδη, ότι όσον αφορά το Αφγανιστάν, βάλαμε ίσω λίγο ψηλά τον πύχη τα πράγματα ήταν περίπλοκα. Σίγουρα κάναμε κάποια λάθη, όλοι μας, όλοι μας. Αλλά προσπαθήσαμε έτσι κι αλλιώς να αλλάξουμε εις βάθος τον τρόπο που θα αντιλαμβάνονται το ίδιο του στο μέλλον οι Αφγανία. Προσοχή. Εμείς οι Δυτικοί είμαστε ανυπόμονη και υπερόπτες πολλές φορές. Και υποχρεώσαμε τη χώρα να εξυγχρονιστεί. Δηλαδή, επιβάλαμε ένα σύνταγμα τρόπο λειτουργίας, μεθόδους, κανόνες κλπ. κλπ. Και τους ήταν ξένο. Δεν έχει καμία σχέση με την ταυτότητα την εθνική με την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους. Δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει από μια χώρα εσαΐ να εξυγχρονίζεται. Σε κάποια φάση θα πρέπει το Αφγανιστάν να ξαναβρει τον εαυτό του, θα πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του και να κρατήσει κάποια στάση ε, εξισορρόπησης. εξισορρόπηση. λέμε Δηλαδή θα πρέπει κάποια πράγματα να έχουν τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, ενώ εμεί κάποια πράγματα του τα επιβάλαμε και λέγοντά του αυτό είναι το σωστό για σας. Ίσως είναι, αλλά ίσω και δεν είναι. Και αυτοί τέλο πάντων να κάνουν τι επιλογέ που επιβάλλονται για το μέλλον του. Και εγώ είμαι πεπισμένο ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τη χώρα αυτή να, να σημειώσει ακόμα μεγάλη πρόοδο. Όχι, θα πρέπει κάπω να κόψουν ταχύτητα. Θα κόψει ταχύτητα και κατόπιν να ανακτήσει αυτή την όθηση, την ορμή προς το μέλλον για την, την, για την διακυβέρνηση, για τη βελτίωση της χώρας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ε, μια, μια μικρή στάση. Γιατί μιλάμε τώρα για, για μια δεκαετία στην οποία συνεχώς έχουμε εξελίξεις και πρόοδο. Και τώρα για να συνεχίσουμε, για τους τη συζήτηση θα πρέπει να μην ξεχνούμε πρόκειται για κυρίαρχη χώρα. Να διέπονται από ερεσιμότητα οι σχέσεις μας με αυτή την κυρίαρχη χώρα. Για να δικαιολογηθεί ο εξομονισμός δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι θα τους προκοδοτούμε εσαΐ να σεβαστούμε την ταυτότητα, να σεβαστούμε τις, τις προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν σε αυτούς τους κανόνες που τους προτείναμε, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να φροντίσουμε να εξαρτάται πάσα οικονομική ενίσχυση από αυτά τα οποία εκεί πρέπει να εφαρμόζονται. Επίσης τώρα, καταπολέμηση ναρκωτικών, διαφθορά, οργάνωση, παιδεία, ε, εκεί, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια προσαρμογής. Ευχαριστώ πάρα πολύ στρατηγέ μου για την περιγραφή αυτή που ξεπερνά τα όρια τα καθαρά της ασφαλείας. Ευχαριστώ, δείξατε πάθος στην περιγραφή. Νομίζω ότι θέσατε το δάχτυλο επί το τύπου των ύλων, επί της διαδικασίας των προβλημάτων της οικοδόμησης κράτους κάτι που ξεπερνά το παράδειγμα του Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν όμως την τελευταία δεκαετία ε, υπήρξε παράδειγμα ακραίο. Ευχαριστώ λοιπόν που συμμεριστήκατε μαζί μας ε, την εμπειρία σας. Νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουμε πολλά από αυτά που είπατε. Μαθήματα λοιπόν είναι αυτά που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, να μας εμπνεύσουν για άλλες περιστάσεις και προβλήματα που εντοπίζουμε και αλλού όπως το κέρας της Αφρικής, στο Σαχέλ, στις περιοχές εκείνες όπου στη θετική εμπλοκή και παρουσία που γίνεται βάση του κατεπήγοντος και νόμιμα και με γνώμονα την αποτελεσματικότητα δεν μας απαλλάσσει από πιο μακροπρόθεσμο προβληματισμό επί της διαδικασίας του nation building. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπερηφανεύεται για τη γενική προσέγγιση, αλλά δεν μπορεί να απαλλαγεί αυτόν τον προβληματισμό. Η μαρτυρία σας λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι άκρως διαφωτιστική. Προφανώς κάποιοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Θέλουν να σχολιάσουν, να σας κάνουν ερωτήσεις. Ο κ. Γκάλερ είναι ο πρώτος. Και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι, σας ευχαριστώ για την ανάπτυξη του θέματος. Νομίζω για το Αφγανιστάν και με όλη την ευρύτητα των θεμάτων που αναπτύξατε πραγματικά μπορώ να πω ότι χρειάζεται χρήση, εκμετάλλευση κάθε δυνατότητα που μας δίδεται. Τα πάντα για τα πάντα. Πράγματι, στους τομείς της παιδείας, της υποδομής και της ασφάλειας μπορούμε να κοιτάξουμε με κάποια υπερηφάνεια τα όσα επιτύχαμε και με τη δική μας υποστήριξη οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των Αφγανών, όπως είπα, που έγινε και με τη δική μας υποστήριξη. Και αυτό είναι το ένα. Βέβαια, του χρόνου θα έχουμε πια το 13ο χρόνο όπου πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή είναι μισή γενιά. δείχνει και αυτό μια θετική εξέλιξη της αφγανικής κοινωνίας. Βέβαια το μέγα θέμα δεν είναι αυτό. Το μέγα θέμα είναι κατά πόσο αρκεί η πολιτική συνένεση μέσα στην ίδια τη χώρα και μετά τη δική μας αποχώρηση για να μπορέσει να συνεχιστεί η προσπάθεια σε αυτούς τους τομείς που ανέφερα. Και εδώ ρωτώ τη γνώμη σας. Καθώς επίσης βέβαια και για την ασφάλεια. θα παραμείνει σταθερή η βούληση των Αφγανών. Είπατε, κύριε, είπατε στρατηγέ μου μάλιστα, μάλλον εσείς, ότι δεν θα καταρρεύσει ο Αφγανικός στρατός. Αυτό το ακούω με μεγάλη ικανοποίηση. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίζονται ορισμένε σημαντικές παράμετροι. Εξού και το ερώτημα. Έχει εξασφαλιστεί στο μεταξύ ότι η αλυσίδα καταβολής των αμοιβών, των μισθών θα διατηρηθεί μήνα τον μήνα ή υπάρχει κίνδυνος να δούμε τελικά τα χρήματα να μην φτάνουν στα χέρια των στρατιωτών. Οπότε τότε πολύ γρήγορα η πίστη τους στο στράτευμα θα εξατμιστεί. Άλλη ερώτηση. Η αποχώρησή μας, η αποχώρηση δηλαδή ε, των διεθνών δυνάμεων Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα γίνει με τρόπο πιο συντονισμένο από ό,τι μέχρι τώρα. Να μην δίνουμε αυτή την εικόνα του τσακιζόμαστε όλοι να φτάσουμε πρώτοι στην πόρτα για να βγούμε. Και τέλος, επειδή μόλις επέστρεψα από το Πακιστάν και μίλησα χθε και με Παστούνους και με τους άλλους, μιλούν για τις εκλογές της 11 μιλούν ταυτόχρονα όμως και για το 2014 και αναμένουν και ελπίζουν και αυτοί να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση. Πόσο έχει προχωρήσει η συνεργασία μας, πόσο έχει προχωρήσει η χρηματοδότηση έργων διαμεθοριακά. Γιατί και από τις δύο πλευρές των συνόρων μπορούν να επωφεληθούν οι άνθρωποι από τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων ώστε ενδεχομένως να συμβάλλει και αυτό σε μια σταθεροποίηση της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά. Uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Είναι πάντα ενθαρρυντικό για μας να ακούμε τέτοια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τέτοια αφοσίωση από τους ειδικού ε, εκπροσώπους και άλλους αξιωματούχους που βρίσκονται σε μια χώρα. Η ερώτησή μου αφορά την απόφαση της Γαλλίας σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Και έτσι εκπληρεί την υπόσχεση να είναι η πρώτη που θα αποχωρήσει από τη χώρα. Αυτό είναι και μια δοκιμή τη ικανότητα των αφγανικών δυνάμεων να επομιστούν τι ευθύνε για την ασφάλεια στη χώρα. Εσεί πώ ε, αξιολογείτε την κατάσταση, Μπορούν οι Αφγανοί να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η απόσυση των Γάλλων, Θα είναι έτοιμοι οι Αφγανοί να επομιστούν την ευθύνη, ή ανησυχείτε για τυχόν εξελίξεις στον τομέα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Οι επικείμενες εκλογές στο Αφγανιστάν. Μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τις εκλογές στη χώρα. Έχουμε ανησυχίες αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νίτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ειδικό μας εκπρόσωπο και τον στρατηγό μας για τις παρουσιάσεις που έκαναν και θεωρώ ότι ήταν αξιοσημείωτη η διορατικότητα και η σαφήνεια της περιγραφής που ε, έβριθε ελπίδες. Πολλά μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε. Ένα από αυτά είναι ότι η διαδικασία της ανοικοδόμησης ή της οικοδόμησης ενός κράτους, μιας χώρας, είναι απείρως πιο περίπλοκο εγχείρημα και πιο μακροχρόνιο από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Όμως ε, δεν πιστεύω ότι πρόκειται επί κινήτρου να μην προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Η συνέπεια να μην το κάνουμε αυτό ε, θα είναι ακόμα χειρότερη. Ακούγοντάς σας πρέπει να πω ότι διαπίστωσα ότι το Αφγανιστάν είναι μια χώρα από τις λίγες που απαγορεύει ο άνδρας μου να επισκεφθώ. Μου λέει ότι είναι αίτιο διαζυγίου. Και μετά από τόσα χρόνια, μη ρωτάτε, τόσο πάνω. Πρέπει να αρκεστώ σε αυτά που μας λέτε. Είχαμε τον Βρετανό Νίκολσον, διπλωμάτης και την γυναίκα του, συγγραφές που ήταν συγγραφές στο τέλος δε, του 30, ήταν στο Αφγανιστάν. Και είχαμε χρήσιμη αλληλογραφία μεταξύ τους, που έδειχνε τις τεράστιες διαφορές πολιτισμικές που υπήρχαν. Κάποια σχόλια ή μάλλον ερωτήσεις. Και οι δύο είπατε ότι πρέπει ότι η ενίσχυση θα συνεχιστεί μετά το 2014 να χορηγηθεί υπό όρου. ερεσιμότητα πρέπει να επικρατεί. Το ακούμε συχνά αυτό. Σας ρωτώ Πώς βλέπετε εσείς την αιρεσιμότητα αυτή. Θα πρέπει να ισχύει για όλη τη χώρα, κατά περιφέρεια, κατά χωριό, κατά επαρχία, κατά πρόγραμμα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς τα βλέπετε, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Αυτή η αιρεσιμότητα, πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Είναι κάπως απογοητευτικό. Έχουμε πολλά προγράμματα στα οποία αναφέρεται αιρεσιμότητα. Αλλά τελικά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς θα εκπληρωθεί αυτή η αδεσιμότητα. Και άλλο ερώτημα που ίσως να είναι προκλητικό. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να εκριζωθεί η καλλιέργεια της παπαρούνας του οποίου και θα είναι και ευκταίο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζέφρι Βαν Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Ζάκας και τον στρατηγό για την υπηρεσία τους στο Αφγανιστάν. Πάρα πολύ δύσκολο μέρος, πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος. Και εκτιμούμε πάρα πολύ ε, τη συνεισφορά σας και σας ευγνωμονούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί θα έλεγα. Ιδιαίτερα σε αυτό το βήμα να μην, να μην συγχαίουμε την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσης με συνεισφορά της ε, ευρύτερης κοινότητας. Αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ ΙΣΑΦ και την ε, πιο ευρία ε, διεθνή κοινότητα και την συνεισφορά αυτού του πλαισίου όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Είναι πολύ πρόημο για να κάνουμε ανάλυση του τι θα ακολουθήσει μετά τις επιχειρήσεις. Εν ευθέτω χρόνο θα λάβει χώρα αυτό. Βέβαια, αρχικός στόχος της ε, παρέμβασής μας στο Αφγανιστάν ήταν να εξασφαλίσουμε ότι το Αφγανιστάν δεν θα ήταν πλέον βάση για διεθνή τρομοκρατία. Ο στόχος πιστεύετε ότι επετεύχθη ή θεωρείτε ότι απλώς μετακινήσαμε και πήγαμε το πρόβλημα δίπλα. Περιγράψατε πολλά καλά πράγματα που κάναμε. Όμως, θεωρείτε ότι ήταν επικοδομητικό να επιβάλλουμε δυτικές πολιτισμικές αξίες σε μια χώρα τέτοια όπως τα Αφγανιστάν. Θεωρείτε ότι αυτό που κάναμε πραγματικά θα διαρκέσει. Και τέλος, μια σκέψη. Σε ποιο στενά πλαίσια η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που απασχολεί. Ποια ήταν τα μεγαλύτερα σφάλματα όσον αφορά την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σύμφωνα με την εμπειρία σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέζιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συχνά λοιπόν άκουσα να μιλείτε για τακτική αποχώρηση στρατευμάτων. Θέλω να θέσω ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στη Γερμανία ακούστηκε πριν λίγο ότι το 2014 θα αποχωρήσουν μεν τα στρατεύματα, θα μείνουν όμως κάποια, κάποια αριθμοί στρατιωτών. Πώς το βλέπετε στο μέλλον, πόσοι συνολικά θα παραμείνουν στη χώρα και επί πόσο διάστημα. Και αυτοί θα έχουν την εντολή μοναχά να εκπαιδεύουν αφγανική αστυνομία και στρατό ή θα προβαίνουν και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Τώρα για την EUPOL μετά το 2014 θα συνεχίσει να εργάζεται η ΕΟΠΟΛ στο Αφγανιστάν. Μιλήσατε και για τον Αφγανικό στρατό και για προβλήματα πληρωμής των στρατιωτικών. Εγώ έρχομαι στο άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα των λιποταξιών, καθώς επίσης και τον μεγάλο αριθμό θυμάτων και στις στρατιωτικές και στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ε, απώλειες διπλασιάστηκαν από το 2011 μέχρι το 2012 βρίσκεται να υπάρχει κάποια εξήγηση εδώ και ίσως να είναι αυτή η αιτία των λιποταξιών και υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για τον αριθμό των λιποτακτών και επίσης για την καλλιέργεια του οποίου το ερώτημα δεν είναι μονάχα αν θα μπορέσει να μειωθεί στην ουσία έχει εκτοξευθεί η παραγωγή του οποίου εκτός από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε παρεμβάσεις σε παρεμβάσεις της Ένωσης ένα ρόλο παίζει πάντα και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθεμπορίου ναρκωτικών. Εσείς θεωρείτε ότι εδώ είναι, πρόκειται για μια ιστορία επιτυχίας. Πώς βλέπετε τέλος πάντων να διαγράφετε το μέλλον και τι κάνετε ώστε να προκαλέσετε εκεί κάποιες αλλαγές. κύριος Αντιπρόεδρος Λίσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής που μπόρεσα να ακούσω τις για την κατάσταση του Αφγανιστάν. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία ήταν θετική και θα θέλαμε όλοι να μοιραστούμε μαζί σας την ελπίδα ότι ο Αφγανικός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν θα μπορέσουν να επομιστούν τις ευθύνες τους για την κάλυψη όλη της χώρας. Αλλά ρωτώ, αν όχι, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν τα καταφέρουν, αν οι συγκρούσει και εμφύλιος πόλεμος στη χώρα επιδεινωθούν, εντατικοποιηθούν περαιτέρω, έχουμε κάποιο σχέδιο ή θα πρέπει κατά την άποψή σα να έχουμε κάποιο σχέδιο για μάχημες δυνάμεις, να επιστρέψουν μάχημες δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Merci, Charles Tannock. Ευχαριστώ, Charles Tannock έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου δεν τον ακούμε δυστυχώς. I too would like to congratulate... Και εγώ θέλω να συγχαρώ και τον ειδικό εκπρόσωπο που θυμάμαι που είχε έρθει για την ε, συνέντευξή του και τον στρατηγό τον ευχαριστώ για το θάρρος τους. Πολύ δύσκολη αποστολή. Ας το χωρίσουμε πάρα πέρα. Αυτό που ανέφερε ο στρατηγός. Κατά πόσο η Δύση υπερφύαλα επέβαλε το μοντέλο της στην κοινωνία του Αφγανιστάν. Παραδοσιακά, στη χώρα μου, κάναμε παρόμοια πράγματα στην Ινδία. Και ήταν μεγάλη επιτυχία. Αφήσαμε κληρονομιά δημοκρατία, κάτω δικαίου και δικαστήρια που δεν υπήρχαν πριν το Ράτζ. Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ιαπωνία επιβάλαμε ένα σύνταγμα. Οι Αμερικάνοι το έκαναν αυτό. Και έσωσαν και τον αυτοκράτορα, που θεωρείται ο εγκληματία πολέμου οι Αμερικοί έδιωξαν ένα βασιλιά που θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο σημαντικό. Τώρα πέθανε, αλλά η βασιλική οικογένεια περιθωριοποιήθηκε. Δίλημα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε την απώλεια αίματος των στατιωτών μας και τα χρήματα που δαπανήθηκαν του φορολογουμένου. Αν βλέπουμε ότι εφαρμόζεται πολύ αυστηρή σαρία, δεν εκπαιδεύονται γυναίκες εκεί. Αντε και γυναίκες καταδικάζονται σε θάνατο, για ομοφιλοφιλία και άλλα ε, πράγματα. Στο εκλογικό μου σώμα. Πώς να τα εξηγήσω. Αν ξαναγίνει μεσονική χώρα σε ένα-δύο χρόνια, επικρατήσει ο φονταμεταλισμό των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, θα με ρωτήσουν γιατί τα κάναμε όλα αυτά, περί σε επρόκειτο. Δηλαδή διώξαμε τα μέλη της Αλκάιντα για να πάνε να συγκροτηθούν στο Μάλι, στην Ιεμένη, στη Σομαλία. Και αυτό που είπε η κυρία Λουέζινγκ. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν κακού ιονού για την παραγωγή οποίου αυξήθηκαν τα η παραγωγή πάνω από 100% παρά την παρουσία ΙΣΑΦ. Και σχετίζεται αυτό με το οργανωμένο έγκλημα, είναι σαφέ. Θα είναι ασφαλέ να αφήσετε πίσω ένα Αφγανιστάν χωρί παρουσία ΙΣΑΦ, που παράγει όλο περισσότερο όπιο και θα γίνει έτσι μια φωλιά για τρομοκρατία και ναρκωτικά. Ίσως η, διαδικασία εκρίζωσης των φυτών και των ναρκωτικών δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ίσως θα μπορούσαμε να αγοράσουμε το όπιο και να το μετατρέψουμε σε φάρμακο. Αντί προτείναμε στους αγρότες να παράγουν ε, είδος τσαγιού, μέντα ή να αλλάξουν την καλλιέργεια και να καλλιεργούν πράγματα με τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν. Και τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το όπιο αυξάνεται. Τώρα που μάλιστα φεύγει το, το ΝΑΤΟ. Αυξάνεται η καλλιέργεια του οποίου. Ευχαριστώ. Ο κ. Σαγκουράκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχω τα, έχω την, τις εξής απορίες ε, με βάση την, την ε, ε, τοποθέτηση κυρίως του στρατηγού de ε, ξέρετε, όταν, όταν έγινε ο, ο πόλεμος ενάντια στο Αφγανιστάν, υπόθηκε ότι η χώρα αυτή ήταν ένα failed state, ένα κράτος το οποίο δεν υπήρχε υποτίθεται. Και ο πόλεμος εκτός των άλλων είχε σκοπό να δημιουργήσει κράτος. State building measures ονομάστηκε τότε. Ο στρατηγός τι γνώμη έχει. Υπάρχει τώρα κράτος. Δεύτερη ερώτηση. Από την τοποθέτησή του με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που εμείς ήμασταν κάθετα αντίθετοι στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, στον πόλεμο στη Ιουκοσλαβία και στον πόλεμο στο Ιράκ και τώρα και στον πόλεμο στο Μάλι. Δεν μπορείς να επιβάλλεις με τη δύναμη των όπλων τον δικό σου πολιτισμό σε άλλους λαούς και πολύ περισσότερο στον 21ο αιώνα. Και δεν έχω την άποψη του κύριου Τάνοκ ότι χάρη στους Βρετανούς οι Ινδοί βρήκανε τη δημοκρατία και βρήκαν το φως, διότι υπήρχαν και άλλοι λαοί που χωρίς τους Βρετανούς βρήκαν τη δημοκρατία και βρήκαν το φως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όμως, έχετε κι εσείς στρατηγέ μου την αίσθηση ότι τα στρατεύματά σας οι Αφγανοί τα θεωρούσαν στρατεύματα κατοχής. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Στρατεύματα κατοχής. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό κιόλας νομίζω, λέτε, ότι δεν μπορούμε να τους εξπολιτήσουμε. Να εξάγουμε τις αξίες της δύση σε μια χώρα. Και άρα είναι μια διαδικασία που πρέπει αυτή η χώρα μόνη της να βρει το δρόμο της. Έτσι είναι. Στρατεύματα κατοχής. Και αν είναι έτσι, δεν νομίζω το πρόβλημα είναι ότι βρήκατε ή ότι το Αφγανιστάν ήταν μια σύνθετη κατάσταση. Ε, το ίδιο αίσθημα μπορεί να υπάρχει και σε άλλε περιπτώσει που είναι λιγότερο σύνθετες οι καταστάσεις και πάλι ο κόσμο να θεωρεί ότι βρίσκεται κάτω από ξένη κατοχή. Ε, τέ, τέταρτο θέμα και τελειώνω με αυτό, ε, μάλλον ε, πρώτο τελευταίο και θα σας πω το τελευταίο ποιο είναι, την άποψή σας την έχουν και άλλοι εγώ σας συγχαίρω για την άποψή σας. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι θα κάνετε με αυτή την άποψη. Καλό είναι να έρθει στη δημοσιότητα. Να ξέρει ο κόσμος. Να ξέρουν, όπως είπατε, οι Ευρωπαίοι πολίτες τι συμβαίνει. Και δυστυχώς σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το κοινοβούλιο σπανίζουν τέτοιες απόψεις. Το αντίθετο υπάρχει. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική. Τελειώνω. Νομίζω ότι ένας από τους πρώην προέδρους της ε, Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα που βέβαια του στήχησε τη θέση του άνθρωπου αυτού. Στην αντιπαράθεση που υπήρχε στη Γερμανία για την παρουσία ή όχι γερμανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, αυτός ο πολύ σοφός άνθρωπος είπε μια μεγάλη αλήθεια. Του είπα, ακούστε κύριοι, τα γερμανικά στρατεύματα πάνε στο Αφγανιστάν για να ανοίξει ο δρόμος για τους Γερμανούς επενδυτές. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, could you please repeat because I, don't got your, question. Παρακαλώ μπορείτε να ε, ε, επαναλάβετε γιατί δεν άκουσα αυτό που το είπατε. Τι λέτε για τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και την ε, τρομοκρατική ενέργεια του Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση από αυτού. Θα σας απαντήσω Μπόστον. Γεια σας. Bien, αυτή αμέσως συζήτηση. Αυτή η συζήτηση. Ας την κάνουμε άλλη μέρα. Άλλη. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα ε, την ισχυτάλη στους ε, προσκεκλημένους μας, στρατηγέ μου, με την αντίστροφη σειρά τώρα. Ε, απαντήστε με ό,τι σειρά θέλετε από τις ερωτήσεις, όποιες ερωτήσεις που έχουν τεθεί θέλετε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αφήσω τα πιο δύσκολα θέματα προς τον πρέσβη, τον κύριο Ζάκας αλλά απαρνιέμαι τον όρο ε, δυνάμεις κατοχής που, δημιουργήσατε, που χρησιμοποίησατε κύριε Βουλευτά, εάν σωστά ερμηνεύτηκε από τους διερμηνείς. δε τον καταγγέλω αυτόν τον όρο, όχι ονόματι της χώρας μου και μόνο που έχασε, τον απορρίπτω. Όχι μόνο ονόματι των Γάλλων και των Βρετανών που πλήρωσαν πολύ υψηλό φόρο αίματος εν των Αμερικανών. Τον απορρίπτω ονόματι των φίλων μας των Αφγανών που δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ οι ίδιοι αυτέ τι λέξει. Αυτέ οι λέξει που θα χρησιμοποιηθούν από ξένου μαχητέ, μάχημε δυνάμει, κυρίω Ταλιμπάν, της Αλ-Κάιντα, που έρχονται να πολεμήσουν στο Αφγανιστάν, αλλά δεν χρησιμοποιείται από του Αφγανούς. Δεν χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από τη φυλή στο Αφγανιστάν. Και ποτέ δεν η παρουσία δυτικών δυνάμεων σαν παρουσία δυνάμεων κατοχής θεωρήθηκαν δυνάμεις αυτούς ότι πραγματοποιούσαν κάποια πράγματα. Όπως πάντα συνέβαινε. Πάντα δεν συνέβαιναν αυτά που επιθυμούσαν. Αλλά δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο κατοχή. Είναι δικαίωμά σα να αναφέρετε τον όρο κατοχή. Δεν τον συμμερίζομαι αυτόν τον όρο και αυτήν την προσέγγιση. Οι Αυγανοί είναι πολύ ευαίσθητοι έναντι τη βοηθεία που του χορηγεί η διεθνή κοινότητα διεθνής κοινότητας για να τους απαλλάξει από ένα φρικτό καθεστώς. Α, αφάνταστο ε, καθεστώς, ένα φρικτό καθεστώς. Χωρίς να σας ε, υπάρχουν εικόνες. Υπάρχει μια ταινία υπέροχη που γυρίστηκε το 2003-2004. Ουσάμα είναι ο τίτλος. Και πήρε βραβείο στις Κάνες, ε, ερμηνείας κλπ είναι τα μικρή κοπέλα, το καθεστώς Ταλιμπάν για να επιβιώσει αναγκαζόταν ε, ε να παντρευτεί με τη βία κλπ. Ε, δεν είναι δικές μας αξίες αυτές. Δεν είναι αξίες μας αυτές. Οι αξίες μας ήταν να βοηθήσουμε να, τη χώρα αυτή, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σεβαστεί την, ε, το να ζουν όλοι μαζί, να σέβεται την ελευθερία, να σέβεται κατά κάποιο τρόπο την ισότητα. Προέχω από μια χώρα που δεν είναι Βρετανική, και εμεί έχουμε κάποιες αδυναμίε στο θέμα αυτό, αλλά σε μια χώρα που αυτές οι αξίες είναι θεμελιώδεις και ουσιαστικές, ουσιώδεις και απετέλεσαν τη βάση πραγματικά των υποχρεώσεων μας έναντι του εξωτερικού ανεξάρτητα από την περιοχή του κόσμου στην οποία έχουμε ε, παρουσία και έχουμε δεσμευτεί. Νομίζω ότι οι Αυγανοί δεν τα βλέπουν έτσι τα πράγματα. Αντίθετα, και εκεί συμφωνώ μαζί σας, ίσως έχουμε εισάγει κάποιε λύσει έτοιμε με το κλειδί στο χέρι. Αυτό προσπάθησα να πω στο Αφγανιστάν γιατί ήταν τα πλούστερο. Τα εργαλεία που ξορίζουμε πολύ καλά, αρκετά περίπλοκα εργαλεία, καμιά φορά πολύ περίπλοκα έναντι της πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα. Και εδώ έγκυται ίσω η δυσκολία και η δυναμία να καταλάβουν οι Αυγανοί. Λένε, να, οι Γάλλοι μας δώσανε μια γαλλική λύση. Οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί. Ε, λειτουργεί σε αυτού, αλλά σε εμά δεν λειτουργεί. Ε, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα διάμεσα στρώματα. Ε, και έχουμε δυσλειτουργία. Διότι ήμασταν κάπω αλαζονικοί, λέγοντα αυτό, αυτό δουλεύει σε εμά, άρα θα δουλέψει και σε εσά. Αντίθετα, στο επίπεδο των αξιών, νομίζω ότι κατάλαβαν πολύ καλά τι μάχη δίνουμε εκεί, ότι η μάχη που δίναμε ήταν μάχη για την ελευθερία, μάχη για την εκπαίδευση των μικρών κοριτσιών, μάχη για να αποφύγουμε τον καταναγκαστικό γάμο, να αποφύγουμε οι γυναίκε να αποκεφαλίζονται, νέε γυναίκε να αποκεφαλίζονται όταν προστατεύει ο πατέρας τους από ε, καταναγκαστικό γάμο να αποκεφαλίζονται. Το 2012, ε, εδώ και τρεις μήνες, ε, και εδώ στάσαμε τη μάχη, το κατάλαβαν. Σε μια συνέντευξη που έδωσα στο, ευρωπαϊκό ραδιόφωνο, γαλλικό ραδιόφωνο, στο Ζαν Πιέρα που είναι πολύ γνωστός στη Γαλλία, ήμασταν δύο που μιλήσαμε και ήταν και μια Αυγανή χειρουργός 40 ετών που την ξέρει ο, ο πρέσβης που είναι χειρούργος η γυναίκα αυτή, που κάθε μέρα πάει στο νοσοκομείο με το φόβο μέσα της, ακόμα και σήμερα. Κάθε μέρα δέχεται απειλέ όταν κάνει την παρέμβασή της, διότι είναι γυναίκα χειρούργος. Είναι πολύ ικανή, είναι καλή χειρούργος. Θέλουν να τους ε, φροντίσει αυτή η γυναίκα. Κάθε μέρα, ε, στο σπίτι και στο νοσοκομείο κινδυνεύει. Έχει απειλέ στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Χωρί και το είπε, πραγματικά εσεί η παρουσία σα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, η παρουσία σα η αμερικανική, η παρουσία των 50 χωρών της συμμαχίας να με κάνουν φοβούμε λιγότερο από πριν. Ακόμα φοβάται προφανώς. Ακόμα υπάρχει δρόμος να περπατήσουν μέχρι να μπορεί να κάνει, ε, να κάνει αυτό που πρέπει χωρίς να φοβάται τι μπορεί να τη συμβεί. Έρχομαι και σε άλλα σημεία που αναφέρθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Η απόσυρση των δυνάμεων. Καταρχά να πω κάτι για τη γαλλική απόσυρση των δυνάμεων, διότι μετέθη το ερώτημα και θα φορέσω το γαλλικό, το γαλλικό μου καπέλο τώρα να απαντήσω στη γαλλική μου ιδιότητα. Η Γαλλία είχε αναπτύξει περίπου 4.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν και είχαμε την ευθύνη κυρίως για μια επαρκία και ένα την επαρχία του Καπισάν και την περιοχή του Ντασιμπή που είναι κοντά στην Καμπούλ ε, και κοντά στον Μπαγκράμ. Όταν ελήφθη η απόφαση να αποσυρθούν οι γαλλικές δυνάμεις Ακόμα και σήμερα περίπου 1.500 Γάλλοι στρατιώτες στο Αφγανιστάν, το υπενθυμίζω αυτό, σήμερα 1.400 περίπου, δεν είναι τα τελευταία στοιχεία, πάνω κάτω. Όταν ελήφθη η απόφαση, η απόφαση ελήφθη από μακρού να επιταχυνθεί η κατάρτιση του τρίτου τάγματος του Αφγανικού στρατού. Εξαρχία και επιταχύνω τις προσπάθειες είχαμε και τύχη να είμαστε εκεί σε μια ζώνη η οποία ήταν λιγότερο βίαιη και λιγότερο κινδύνευα από άλλες. Δεν είναι η πιο... Ε, ε, ε, δεν είναι πιο επικίνδυνη περιοχή, Σαμντίμ και αλλού, Ασανγκάρ, Καζακή κλπ. Είναι περιοχές που είναι πολύ πιο επικίνδυνες και η αντίσταση των Ταλιμπάν είναι πολύ πιο καλά εμπεδωμένη και δρεωμένη. Στο Καπισάν δεν ισχύει αυτό στην επαρχία. Έπρεπε εκεί να έχουμε προβάλλουμε αντίσταση που ήταν όμως στις δυνατότητες των Αφγανών. Αποσύραμε δυνάμεις, τις μάχημες δυνάμεις, οι τελευταίοι φύγαν το μήνα Νοέμβριο, Έκτοτε οι Αυγανοί έχουν αναλάβει την ευθύνη της περιοχής που ήταν υπό την ε, γαλλική εποπτεία. Από ό,τι γνωρίζω, οι Ταλιμπάν δεν ξανακέρδισαν ούτε εκατοστό εδάφους. Αυτό δείχνει ότι οι δυνάμει ασφαλεία εκεί, σε αυτά τα κομμάτια, δεν είναι παντού τα ίδια τα πράγματα στο Αφγανιστάν. Πάντω οι δυνάμει εκεί μπορούν να αντιμετωπίσουν τι ευθύνε του. Ο κυβερνήτη Σαφίκ του Καπιστάν, ο στρατηγό ε, του Τρίτου Τάγματο, του ΦΟΠ και λοιπά και των Εθνικών Δυνάμεων του Αφγανιστάν, όλοι οι διοικητέ και τη αστυνομία, όλοι είπαν οι αρμόδιοι ότι έκαναν, τα καταφέρουμε, τα καταφέρουμε και τα κατάφεραν. Και πιστεύω ότι αυτό το μικρό κομμάτι του Αφγανιστάν, μικρό κομμάτι, δεν είναι πολύ μεγάλο τμήμα, δεν θα πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν. Αντίθετα υπάρχουν πολλά προβλήματα διακυβέρνησης και προβλήματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Όσον αφορά το συντονισμό της απόσυρσης των δυνάμεων, μου ετέθη ένα ερώτημα όσον αφορά το συντονισμό τη απόσυρση των δυνάμεων, πώ οργανώνεται, είναι μία από τι ευθύνε μου. Είναι πραγματικά οργανωμένη η απόσυρση. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε και προβλήματα, πραγματικά προβλήματα. Ε, είμαστε έχουμε τα σύνορα με το Πακιστάν που είναι κλειστά. Είναι εσόκλειστη η χώρα. Δεν φύγαμε μέσω του Ιράν. Έχουμε τα σύνορα με το Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, τα Ταϊστάν στο βορρά που έθεσαν και θέτουν ακόμα προβλήματα σημαντικά. Λοιπόν, η απόσυση των δυνάμεων για τους Αμερικανούς βασικά, επιθυμίζω ότι οι Αμερικανοί αρχίσαν να αποσύρουν το 2011 10.000 άντρε που ε, έφυγαν το τέλο του 2011, απέσυραν 23.000 άντρε το 2012. Ταυτόχρονα εμείς οι Γάλλοι αποσύραμε 2.500 άντρε, οι Βρετανοί απέσυραν 500-600 άντρες, οι Γερμανοί 500, 600 αντρε οι γερμανοι 500 οι ισπανοι κλπ. κλπ. Από μνήμη τα λέω αυτά. Εκενώσαμε και αποσύραμε τους άντρε μας για ε, τις εναερίου οδού δεν σας εκπλήσει αυτό. Αλλά ο εξοπλισμός βγαίνει ε, από τις ενεργείες οδού. Είτε με άμεσες πτήσεις προς τις χώρες προέλευσης για το πιο ευαίσθητο υλικό, είτε με πτήση προς χώρες του κόλπου και εκεί πάμε φορτώνουμε στα πλοία προς τη ΣΥΠΑ, προς τη Βρετανία, ε, προς την Ευρώπη. Βρετανία, Ευρώπη όταν μιλώ για τις άλλες χώρες. Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Και η μάχη ακόμα εκεί είναι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, για το συντονισμό. Ε, δεν, είδα, δεν είδα κάποια ταξία, άτακτη απόσυρση. Ίσως κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια συντονισμού της απόσυρσης των δυνάμεών μας ε, τι διάφορε μονάδε, λαμβάνοντα υπόψη και των διάφορων χωρών, λαμβάνοντα υπόψη τις ευαισθησίε και τι ανάγκε εθνικέ, τι ανάγκε επιτόπιε, την παρουσία των Αφγανών να μην φύγουμε πιο νωρί και αν φεύγαμε πιο νωρί από ό,τι είχαμε ε, υπολογίσει όταν κάναμε το assessment, την αξιολόγηση, τα πράγματα καλά πήγαν, καλά συντονίστηκαν, αντιμετωπίσαμε προβλήματα που αφορούσαν τα κλειστά σύνορα. Άρα η εκένωση αυτή ουσιαστικά γίνεται δια της εναερίας οδού και είναι πολύ δαπανηρή. Αν ανοίξει σύνορο με το Πακιστάν, ε, κάναμε κάποια διαβήματα, Υπάρχει ο κίνδυνος επίθεσης πάντα στο έδαφος του Πακιστάν και είναι από τους μεγάλους φόβους αυτό των Πακιστανών. Δηλαδή, να τους δαχτυλοδείξουμε ότι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν ε, τις ε, δυνάμεις του ΟΤΑΝ που εκενώνουν προς το Καράτσι. Από Να πληγούν από εσωτερικέ μάχε πάνω στο έδαφο του Πακιστάν, Ξέροντα ότι η ευθύνη για τι δυνάμει, για την εφοδιοπομπή, για τι δυνάμει, ε, είναι στα χέρια των πακιστατικών δυνάμεων και είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα για το Πακιστάν. Και μπορούμε να το καταλάβουμε το φόβο του Πακιστάν. Τώρα, όσον αφορά τη βάση για τρομοκρατία, αν θα ξαναγίνει η βάση μια μέρα, το, το Αφγανιστάν ξανά για, τις, για τους τρομοκράτες. Εκριζώσαμε την Αλκάιντα στο Αφγανιστάν. Την εκριζώσαμε, την εξαλείψαμε. Πάει. Τι σημαίνει εκριζώνω. Τους διώξαμε, τους κυνηγήσαμε. Τους παρατηρήσαμε, παρακολουθήσαμε, τους εξουδετερώσαμε, τους συλλάβαμε. Σε διάφορες περιοχές, την άνοιξη του 2012, το Τουνάρ και το, το καλοκαίρι του 2012, οι επιχειρήσεις μας στέφθηκαν από επιτυχία. Και είδαμε κάποιους ξένους μαχητές που ήρθαν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν. Χτυπήθηκαν σκληρά από άκρο αποδοτικά μέσα που χρησιμοποίησαμε και του είδαμε να φεύγουν, να αποσύρονται. Πηγαίνοντα προ άλλε περιοχέ όπου μπορούσαν αυτοί ε, να κάνουν τι κακέ του πράξει. Του ακούσαμε να φεύγουν, του είδαμε να φεύγουν, του παρακολουθήσαμε στην αναχώρησή του. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλε περιοχέ του κόσμου όπου αυτοί οι μαχητές σήμερα μπορούν να δράσουν και να δράσουν κατά των συμφερόντων μας ή τουλάχιστον να αποσταθεροποιήσει τα συμφέροντά μα. Τώρα γυρίσουμε στο Αφγανιστάν. Δεν υπάρχουν πια στο Αφγανιστάν. Θα γυρίσουν ξανά αυτοί στο Αφγανιστάν. Όχι. Αυτή που είναι περιθωριακή η παρουσία του στο Αφγανιστάν. Σχεδόν δεν μπορεί να εντοπιστεί. Θα επανέλθουν. Ναι. Αν είναι rogue state, αποτυχημένο κράτο, failed state, που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει σαν χώρα το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει παντού. Παντού ισχύει το ίδιο. Το Αφγανιστάν από αυτή την έποψη δεν διαφέρει από μια άλλη χώρα δεν είναι διαφορετικό, διαφορετική από το Σαχέλ, από τη Σομαλία, από το Σουδάν, από τη Συρία, από την Ιεμένη. Το διακύβευμα για να μην ξαναγίνει βάση το Αφγανιστάν για τη διεθνή τρομοκρατία είναι το αφγανικό κράτος να έχει τα ελάχιστα μέσα να μπορεί να επιβάλλει τη διακυβέρνηση και να επιβάλλει τους όρους ασφαλείας. Αν κατατύχει αυτό δεν πραγματοποιηθεί, φυσικά διότι η φύση γεμίζει το κενό, οι μαχητές οι Ισλαμιστές θα επανέλθουν, θα εγκατασταθούν ξανά στις περιοχές εκείνες ε, που μπορούν να κινηθούν ατιμωρητοί. Αλλά δεν μπορούμε να προβούμε σε μια τέτοια αξιολόγηση τώρα όσον αφορά το θέμα. Όσον αφορά τι γίνεται μετά το 2014, ετέθη το ερώτημα τι θα συμβεί μετά το 2014. Μετά το 2014 αποφασίστηκε να παραμείνουν δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Resolute Support είναι η αποστολή του ΝΑΤΟ μετά το ISAF 2014 που θα παραμείνει στο Αφγανιστάν. Και αυτή η αποστολή υπό εντολή του ΝΑΤΟ ε, δεν θα είναι αποστολή μαχήμων δυνάμεων αλλά θα είναι για την ε, κατάρτιση, συνεχή κατάρτιση ε, μεταδόση τεχνογνωσίας, εκπαίδευση διδασκαλία στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν, δυνάμεις εθνικές ασφαλείας του Αφγανιστάν, που θα αναλάβουν τη μάχη αυτές. Κυρία μου, είπατε ότι αυτές οι εθνικές αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας είδαν απώλειες στις μάχες, να διπλασιάζονται οι απώλειες στη μάχη. Δεν χρησιμοποιήσατε απόλυτα αυτόν τον όρο. Μεταξύ 2011-2012. Ναι, διότι όλο και περισσότερο αναλαμβάνουν ευθύνες και πράγματι ε, αυτές αρχίζουν να μάχονται. Ενώ εμείς αρχίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας και να περνάμε σε μια θέση υποστήριξης των δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Και αν βλέπατε τα στοιχεία, τις απώλειες που έχουμε υποστεί στο ISAF από το 2011 με το 2012, από ό,τι θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, όσον αφορά κάποιες μονάδες, χάσαμε πάνω από 520 στρατιώτες το 2011 και 300 το 2012. Σχεδόν το μισή, μισό από τις λιγότερο, λιγότερες απώλειες από ΙΣΑΦ και πάλι είναι πολύ. Ε, σημαντικές απώλειες. Δηλαδή είναι βία οι μάχες, αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν ηγούνται, όχι ακόμα παντού, αλλά σε πολλές περιοχές και ηγούνται, επομίζονται τις ευθύνες τους που συνδέονται με την ειρήνευση και σταθεροποίηση της χώρας έναντι των ε, δυνάμεων αυτών ε, των ε, προσπαθούν να ανατρέψουν το νόμιμο καθεστώ και να επιβληθούν. Αυτά έχω να πω στι διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν κυρίως στα στρατιωτικά θέματα, να πω μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά τα ναρκωτικά. Πρώτα απ' όλα τα ναρκωτικά κάνουμε καθημερινή μάχη γι' αυτό. Αμερικανοβρετανική κυρίως, με αποτελέσματα έξοχα εξαιρετικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πολεμάμε. Υπάρχει μια task force αμερικανοβρετανική που δεσμεύτηκε να κάνει τη μάχη κατά των ναρκωτικών. Ακόμα και αν σε άλλες χώρες, από άλλες χώρες υπάρχει συμμετοχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι, είναι ε, μικρά. Νομίζω τα αποτελέσματα είναι ε, πράγματι ενθαρρυντικά. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ότι έχουμε πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των δικτύων των ναρκωτικών, των εγκληματικών δικτύων, των δικτύων των Ταλίμπαν και των πολιτικών δικτύων. Διασυνδέονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αν πούμε κάτι άλλο θα ήταν ψέμα. Και δεν συνηθίζω να ψεύδομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Πρέπει να επιτεθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Προφανώ, όταν λέμε πρέπει να επιτεθούμε στο πρόβλημα, όλοι σηκώνουν τα χέρια στον ουρανό και λένε Ω Θεέ μου, είναι αδύνατον. Αλλά τι έκανε ο πρόεδρο Ερίμπε στην Κολομβία μεταξύ 2002 και 2007. Καταπολέμησε του ΦΑΡΚ, τα κατάφερε. κατα... Τα δίκτυα ναρκωτικών στην Κολομβία τα κατάφερε. Αναδιοργάνωση πλήρης του κρατικού μηχανισμού της Κολομβίας ούτω ώστε να εκριζωθεί πραγματικά και το ναρκωτικό και η ΦΑΡΚ. Μεταξύ, μεταξύ από εσά, μετα, με, με, μερικοί από εσά ε, ξέρετε καλύτερα και ήμουνα 15 μέρες τόπου εκεί. Ε, υπήρχε μεγάλη υποστήριξη στο μεγάλο σύμμαχο των Αμερικανών που έδινε πληροφορίες και μέσα και, και εκπαίδευση για να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει δυνάμεις. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε ε, από αυτά που συνέβησαν στην Κολομβία. Βλέπουμε ότι η πολιτική βούληση, μια κρατική οργάνωση που απορρέει από αυτή και μια διεθνής βοήθεια πραγματική, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Αφγανούς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους, να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα αυτά που είναι σαν τα πόδια δικτυωμένα ε, για να πετύχουν αποτελέσματα. Και όσο πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. 2008, 2009, 2010 τα πραγματικά αποτελέσματα εδώ και τέσσερα χρόνια τα είδαμε στο Αφγανιστάν το συζητήσαμε με του Αφγανού φίλου μα το, το πρόβλημα αυτό, τον Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Αμήνε και με τι υπηρεσίε καταπολέμηση των ναρκωτικών που είναι αποτελεσματικέ. Αντιμετωπίζουν όμω αυτά τα τέσσερα δίκτυα που προανέφερα. Τα κυκλώματα και θα πρέπει να, να πάρουμε μαθήματα όσον αφορά την οργάνωση, την πολιτική βούληση και μαθήματα όσον αφορά τη διεθνή υποστήριξη, ούτω ώστε αποτελεσματικά να καταφέρουμε να εκριζωστεί αυτή η απειλή που είναι απειλή άμεση κατά των συμφερόντων μα και των αξιών μα. Σα euh, Σας ευχαριστώ, στρατηγέ. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από τις εκτεταμένες απαντήσεις του αγαπητού στρατηγού, είμαι πολύ πιο χαλαρός εγώ τώρα για να μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που παραμένουν ίσως αναπάντητες. Πρώτα για το θεμελιώδες αυτό ερώτημα, δηλαδή εάν έχουν επιτευχθεί οι αντικειμενικοί στόχοι της διεθνούς παρέμβασης. Ναι για την ώρα. Αυτό θα απαντήσω. Είναι σαφής η πρόοδος και ορατή, αλλά είναι και εύθραστη. Και για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας, την παροχή υποστήριξης προς τη χώρα αυτή, βέβαια με όλο το σεβασμό των παραδόσεων και θύμων κλπ. Ανοίγει αυτή τη φορά, αυτή, ανοίγει αυτή τη στιγμή, ανοίγει και σε ό,τι αφορά τις αρχές και τις αξίες. Όταν μιλούμε για αλαζονία, για την επιβολή των δικών μας συστημάτων αξιών κλπ. Αυτό πρέπει να το αντισταθμίσουμε και με την επιθυμία, τις επιθυμίες των ανθρώπων των ίδιων στη ρίζα της χώρας αυτής. Όταν πήγα εγώ να παρακολουθήσω τη ψηφοφορία στις εκλογές ουρές ανδρών και γυναικών παρά τις απειλές των Ταλιμπάν. Η περηφάνεια που έδειξαν όταν πήγαν να ρίξουν την ψήφο τους. Οι αριθμοί των παιδιών που πάνε τώρα στο σχολείο και που δείχνει και πόσο κρίσιμη είναι η εκπαίδευση και για αυτούς είναι πραγματικά έμπνευση για μας. Ένα τώρα βέβαια από τα διδάγματα που οφείλει να συναγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Αμερικανοί και οι άλλοι διεθνεί μας εταιρείοι είναι ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέμε quick fix, δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις. Και ο στρατός δεν μπορεί μόνος του να ανταποκριθεί. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα εκεί και στις περιοχές συγκρούσεων αλλά και στην περίοδο μετά την σύγκρουση. Δηλαδή χρειάζεται και η capacity building και να δημιουργηθεί δηλαδή ικανότητα για να σταθεί η χώρα στα πόδια της και η οικονομική ανάπτυξη. Και βεβαίως μέσα σε πλαίσιο σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με την ευρύτερη έννοια. Υπάρχει, με ρωτάτε, πολιτική συνένεση σε ό,τι αφορά την διατήρηση αυτών των επιτευμάτων. Εγώ βλέπω θετικές εξελίξεις. κάποιος από τους ευρωβουλευτές με ερώτησε σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις, στο Αφγανιστάν. Εγώ θυμάμαι πολύ καθαρά τις πρώτες μου συζητήσεις με πρώην Αφγανούς ηγέτες προτριετίας όπως τον Μουλάζα είναι και άλλους Τα μιλήσαμε για δικαιώματα των γυναικών η απάντησή τους ήταν απορριπτική, αλαζονική μου είπανε τι μας μιλάτε εδώ για δικαιώματα των γυναικών. Αυτές που έρχονται εδώ και μιλάνε για δικαιώματα μου είπαν. Δεν είναι Αφγανές. Αυτές τις έχουν πληρώσει οι Αμερικανοί για να έρθουν εδώ να μας πούνε και να σας πούνε αυτά που θέλουν οι ίδιοι. Και όμως είχαμε 80 κορίτσια μεταξύ των πρώτων 400 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Καμπούλ. Αρχίζει λοιπόν και αλλάζει η νοοτροπία. ο Ραχατζάν Μουτασίμ που έχει εκδώσει δήλωση τελευταία και που έχει δηλώσει ότι προτίθεται να σχηματίσει πολιτικό κόμμα και λέει καθαρά και δημόσια ότι υποστηρίζει και εκτιμά τις αλλαγές που επέφερε η, η διεθνής κοινότητα και για την πρόοδο και για την εκπαίδευση και στα δικαιώματα των γυναικών. Δεν θα έλεγα ότι έχει πραγματικά θεμελιωθεί μια πολιτική συνένεση. Υπάρχει όμως μια μετακίνηση προς μια βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στο Αφγανιστάν, προς μια καλύτερη διακυβέρνηση και, και μια πιο έντονη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών που έχει αυξηθεί στη χώρα. Αυτά τα επιτεύγματα, όπως είπα, εξακολουθούν να είναι εύθραστα. Και για το λόγο αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη, αλλά με όρους. Η κυρία Κοπά με ρώτησε, όχι με συγχωρείτε, η κυρία Νέιτς, με ρώτησε για την αιρεσιμότητα, για τους όρους δηλαδή. Αν γίνεται αναπεριφέρεια, αναέργο ή συνολικά στη χώρα. Η κυβέρνηση ε, του Αφγανιστάν πρώτα πρέπει να επιβάλλει όρους. Εάν θέλουμε εδαφική ακαιρεότητα, έχουμε πρώτα-πρώτα απέναντί μας την κεντρική αφγανική κυβέρνηση. Με την παροχή διευκολύνσεων σε αυτούς, με την βοήθεια που τους προσφέρουμε για να θεσπερίσουν τις ελευθερίες στην, ε, ε, σε όλη την επικράτεια, αλλά ταυτόχρονα καθιστώντα τους υπόλογους και απέναντι στους πολίτες και απέναντι στους δωρητές. Γι' αυτό και μιλούμε για την αρχιτεκτονική της αιρεσιμότητας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που έδειξε τη σοβαρότητα τη στήριξη των κανόνων του παιχνιδιού και ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει μετά από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε όλοι μαζί στο Τόκιο. Και αυτό απασχολεί όλους και στις Βρυξέλλες αλλά και τις χώρες μέλη, βεβαίως και την Ουάσιγκτον. Σε ό,τι αφορά τις επικείμενες εκλογές, αν έχουμε ανησυχίες. Ναι, βεβαίως έχουμε ανησυχίες όπως και τα παλαιότερα χρόνια. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δυστυχώς αποτύχαμε να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθεί στο Αφγανιστάν ένα αξιόπιστο σύστημα ε, καταγραφής των ε, ε, ψηφοφόρων. Έχουμε ακόμα τμήματα του Αφγανιστάν τα οποία δεν καλύπτονται και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με την Αφγανική κυβέρνηση και με την κοινωνία των πολιτών. Βέβαια, το θετικό σημείο είναι ότι τούτη τη φορά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη οριμότητα. Το βλέπουμε στις συζητήσεις μεταξύ των Αφγανών φορέων, των Αφγανών stakeholder. Το 2014 δεν είναι ακόμα μια χρονιά εκλογών, είναι μια πραγματική χρονιά μεταφοράς των ευθυνών στους ίδιους τους Αφγανούς. Και γι' αυτό χαιρόμαστε και για τη συζήτηση την οποία διεξάγουν μεταξύ τους για την στερέωση, θεμελίωση ε, πολιτικών κινημάτων, δημιουργία κομμάτων. Επίσης, ο πρόεδρος Καρζάη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συνδιαλλαγής με νέους επιτρόπους. Η νομοθεσία παίρνει το δρόμο της, λαμβάνει μορφή σιγά σιγά μέσα στην Αφγανική Ζήργα, το, τη Βουλή θα γίνουν εκλογές όχι όπως ίσως αυτές που βλέπετε στην Ελλάδα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού, αλλά πιστεύω ότι θα έχουν περισσότερη κυριαρχία ήδη Αφγανοί, την ownership που λέμε, και ένα αποτέλεσμα που θα γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των Αφγανών. Είναι δυνατό και επιθυμητό να ξεριζωθεί η καλλιέργεια του οποίου στο Αφγανιστάν. Ναι, είναι δυνατόν, είναι επιθυμητό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι εξακολουθεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος για τους Ταλιμπάν, διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, ολιστικά όπως λέμε, και αυτό είναι που επίμονα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και για την ε, φύλαξη των συνόρων και, και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη και την προσπάθεια να προσφέρει άλλες πηγές εισοδήματο. Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να γίνει και από την πλευρά των χωρών που εισάγουν τα ναρκωτικά. Πρέπει να γίνει και αυτή η συζήτηση, δηλαδή πώς να αντιμετωπιστεί η κατανάλωση. Αυτό βέβαια ξεφεύγει από τα όρια της ε, αρμοδιότητας και της εντολής μου. Είναι δική σας εντολή και δική σας αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά είπα για άλλα θέματα. Ο κύριος Λίσεκ με ρώτησε εάν... Α, έχει αποχωρήσει από ό,τι βλέπω. Αλλά ίσως κάποιος μπορεί να του μεταφέρει την απάντησή μου για την αποχώρηση των δυνάμεων. Το χρονοδιάγραμμα της αποχωρήσεως έχει καθοριστεί πλέον σαφώς. οι στρατιωτικές δυνάμεις θα μειώσουν σημαντικά την παρουσία τους από το 2014. Οφείλουμε να σεβαστούμε την κυριαρχία του Αφγανιστάν και ταυτόχρονα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν οι ίδιοι να διατηρήσουν την ασφάλεια αλλά και την τάξη μέσα στη χώρα τους. Εν τέλει, επιθυμώ να σας ευχαριστήσω. Υποστηρίζω τις θαυμάσεις απαντήσεις που σας έδωσε ο στρατηγός σας ευχαριστώ όλες και όλους για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον που δείχνετε για το Αφγανιστάν. Χώρα η οποία πέρασε παραπάνω από 30 χρόνια πολέμου και συγκρούσεων και που αξίζει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χώρων μελών της. Τα δικά μου καθήκοντα λήγουν την 1η Σεπτεμβρίου. Ελπίζω εσείς ωστόσο να συνεχίσετε την δέσμευση και το ενδιαφέρον σας στο Αφγανιστάν και να προσφέρετε την απαραίτητη υποστήριξη, βεβαίω και χρηματοδοτικά, μέσα στη νέα δημοσιονομική σας προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, κύριε μάλλον στατηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την μαρτυρία σας. Ήταν πάρα πολύ ποιοτική η παρουσίασή σας. Ξεπεράσαμε μια απλή καταγραφή της καταστάσεως, απλή διαπίστωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Είδατε κατά τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι αυτό ένιωσαν. Κύριε Πρέσβη, έχετε διάφορα αιτήματα σας κάναμε ε, απέναντί μας, κυρίως δημοσιονομικής φύσεως. Βοηθήστε μας κι εσείς να κάνουμε, ετοιμάσουμε αυτή την αποστολή κοινοβουλευτική στο Αφγανιστάν. Ξέρετε το θέμα, αυτή η υποεπιτροπή θεωρεί ότι επί, μακρόν ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Αφγανιστάν και ποια μεγαλύτερη απόδειξη ενδιαφέροντος από το να πάμε επί τόπου. Με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο να υλοποιήσουμε αυτή την αντιπροσωπεία, την αποστολή μας, την αρνούνται για λόγους ασφαλείας κάθε χρόνο, παρόλο που οι συνάδελφοι μας εθνικών κοινοβουλίων κάνουν πολύ συχνά επισκέψεις στο Αφγανιστάν χωρίς πρόβλημα. Χάρη σε εσά ε, προχωρήσαμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο επίσκεψη πάντα τον, ε, το φθινόπωρο. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα ε, στη συνεδρία των επικεφαλής αντιπροσωπιών. Για και εκείνοι είχαν έρθει στην Επιτροπή μας, οπότε μην διστάσετε. Make the point. Να, να, να απευθυνθείτε σε εμά εδώ στι Βρυξέλλε, στο Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε επί τόπου να τα πούμε. Ε, Σα το στρατηγό, δεν ξέρω να συνδέσουμε δυστυχώ, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, σημαντικά όσα μας είπατε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ το χρόνο που μας διαθέσατε και για την ανοιχτή σας στάση κατά τη συζήτησή μας. Συνάδελφοι, ευχαριστώ που ήρθατε. Θα σας υπενθυμίζω ότι αύριο θα συνεχίσουμε στις 9.30 και έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροπλάνα drone. Ευχαριστώ.